Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινήσουμε σιγά σιγά την ε, ακρόασή μα. Λοιπόν. Και μετά θα ξεκινήσουμε και μια συζήτηση με του ε, σκιώδε ηγητέ που είναι παρόντες. Και με συγχωρείτε για την ε, καθυστέρηση. Κύριε Ντεπρέ, παρακαλώ, ξεκινήστε. Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητέ Κλοντ, δεχτεί η συγγνώμη σας. Και εγώ το πρωί, προβλεπόμουν το πρωί και δεν ήμουν παρόν. Ευχαριστώ που δεχτήκατε λοιπόν να αναβληθεί η παρουσίασή μου κατόπιν ετοιματός μου για το απόγευμα. Κύριε Πρόεδρε, ποιο είναι το θέμα μας. Πρόκειται για ένα σχέδιο κανονισμού με στόχο την εναρμόνιση των στοιχείων ασφάλειας, ε, των ταυτοτήτων ε, και των ε, καρτών διαμονής για τους επικόους που διαμένουν, μάλλον για τους διαμένοντες στην Ένωση και για τα μέλη της οικογένειάς τους. Ποιος είναι ο στόχος, πρέπει να είναι ξεκάθαρος για όλους μας, είναι πάνω και πρώτα απ' όλα η διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων ελεύθερης διακίνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως γνωρίζετε, η Ευρώπη κυκλοφορούν μεταξύ των διαφόρων χώρων της Ένωσης. Έχουμε 15 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες που διαμένουν σε άλλο κράτος με μέλο από αυτό στο οποίο κατάγονται και εκ των οποίων 11 εκατομμύρια εργάζονται κιόλα σε ένα άλλο κράτο μέλο. Για να τα πω πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Ο στόχο δεν είναι η αντικατάσταση των δελτίων ταυτότητα των εθνικών ταυτότητων με μια ευρωπαϊκή ταυτότητα. Παραμένουν εθνικές οι ταυτότητες. Ούτε τίθεται θέμα να υποχρεωθούν τα κράτη-μέλη που δεν έχουν να δίνουν ταυτότητες αν δεν τις εκδίδουν, δεν θα υποχρεωθούν να το πράξω. Στόχο είναι εναρμόνιση των στοιχείων ασφαλείας, των χαρακτηριστικών ασφαλείας των δελτίων ταυτότητας που έχουν τέτοια. Ποια είναι τα στοιχεία που προτείνω να συμπεριληφθούν όσοι συμπληρωματικά στοιχεία των διατάξεων της Κομισιόν. Και λέω ξεκάθαρα ότι θέλεις να λάβω στο μέγιστο βαθμό υπόψη μου τις ε, συστάσεις ε, του ΦΡΑ ε, και του επόπτη δεδομένου. Διάβασα επίσης την, Επιτροπή, την έκθεση Επιτροπής Γυναικών και τις συστάσεις ό,τι αφορά τη διάσταση του φύλου. Αυτό που ζητώ λοιπόν πρώτα απ' όλα είναι στον κανονισμό αυτό να διευκρινιστεί ότι δεν αποτελεί νομική βάση για τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Τράπεζας Βιομετρικών Δεδομένων. Γιατί ξέρω ότι ορισμένες πολιτικές ομάδες έχουν αυτήν την ανησυχία, τα λέω ξεκάθαρα λοιπόν, απόλυτα ξεκάθαρα και εξού περιέλαβα και το σημείο αυτό στο, στην έκθεσή μου. Δεύτερο δεν θα χρησιμοποιηθεί ο κανονισμός αυτός ως νομική βάση από κάποιο κράτος μέλος για να συγκροτήσει Εθνική Τράπεζα Βιομετρικών Δεδομένων αν θέλουν να το κάνουν αυτό κάποια κράτη-μέλη, δεν θα μπορέσουν να το κάνουν βασιζόμενα πάνω σε αυτόν τον κανονισμό. Δεν είναι νομική βάση ο κανονισμός για κάτι τέτοιο. Αυτές είναι πρώτες διευκρινήσεις που θέτω υπόψε. Δεύτερον, θέλησα να ενισχύσω τις εγγύησεις για τον τρόπο με τον οποίο τα βεντρικά δεδομένα θα συλλέγονται και ιδίω όταν μιλάμε για παιδιά ή για ευάλωτα άτομα. Δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες. Προβλέπω όμως συγκεκριμένε εγγύησεις, πέραν αυτών που είχαν περιληφθεί στην αρχική πρόταση. Τρίτον, συμπληρώνω κάποια κενά κατά την απόψή μου στην πρόταση, στο αρχικό κύμα της Κομισιόν, σε σχέση με την προστασία δεδομένων. Ρητός προβλέπω τα δεδομένα να διατηρούνται από τη στιγμή που έχουν συλλεγεί εκτός του τσίπ μόνο ε, όσο διαρκεί η ισχύ της άδεια ε, και για ένα μήνα μετά από τη λήξη. Όταν θα έχουν συλλεγεί και ενσωματωθεί στο τσίπ ε, τα δεδομένα πρέπει να καταστρέφονται. Προβλέπω επίσης διατάξεις για να περιοριστεί η χρήση των βιομετρικών δεδομένων, ώστε να μην μπορεί να γίνει χρήση τους από ιδιώτες ή ιδιωτικές υπηρεσίες. Εκτός σε σχέση με ό,τι προβλέπεται ρητός σε ό,τι την μεταβίβαση των αρχικών δεδομένων στην, στο τσίπ. Προσθέτω επίσης μια διάταξη, η οποία προβλέπει πολύ ξεκάθαρα ότι τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για την ε, καλή επεξεργασία ε, των δεδομένων με βάση τον κοινωνικό κανονισμό για την ε, ασφάλεια των δεδομένων. Και όταν ε, απευθύνονται σε ξένες υπηρεσίε εκτός του ιδιωτικού τομέα, για την ταυτότητα, για την παραγωγή της ταυτότητας. Και προσθέτω και μία ιδιαίτερη διάταξη ξεκάθαρη που λέει ότι όλα τα κράτη-μέλη αναγνωρίζουν μεταξύ τους το δελτίο ταυτότητας ως έγγραφο ταυτότητα και ταξιδιωτικό έγγραφο για να μην υπάρχει αμφισβήτηση. Επίση προβλέπω και αυτή η διάταξη δεν υπήρχε στο αρχικό κείμενο. Θα σας δώσω κάποιε λεπτομέρειε. Η διάταξη λοιπόν υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να ανταλλάσσουν μεταξύ τους τι κλίδε κλίδες των βιομετρικών δεδομένων. Εξεργαζόμαστε σε αυτό το φάκελο είδα ότι τα βιομετρικά δεδομένα που έχουμε στα διαβατήρια Μπορεί να τα διαβάσουν μόνο ε, το, το κράτος μπορεί να τα διαβάσει που έχει εκδώσει το διαβατήριο και όχι τα άλλα. Δεν μπορούμε να στήσουμε 370-400 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες να δώσουν γενικά δεδομένα τα οποία μπορεί να τα χρησιμοποιεί μόνο η χώρα ε, που το έχει εκδώσει το διαβατήριο και όχι να μην έχουν πρόσβαση υπηρεσίες ασφαλείας ή τα ε, οι συνοριακές αρχές. Γιατί έτσι χάνει ε, μέρος της, του λόγου ύπαρξής του το έγγραφο αυτό, το διαβατήριο. Επίσης, προβλέπω με κάποιες άλλες διατάξεις να εμποδιστούν τα κράτη-μέλη, μάλλον να μην βρεθούν τα κράτη-μέλη απέναντι σε μεγάλο φόρτο για την αντικατάσταση των φυστάμενων ε, ταυτοτήτων και να τις αντικαταστήσουν δηλαδή με άλλες καινούριες. Ζητώ επίση από την Κομισιόν τα κρατημέλη να αναπτύξουν καλύτερε πρακτικές σε ό,τι αφορά το αρχικό κείμενο, το πηγαίο έγγραφο, source document. Να υπάρχουν επίση προσωρινά έγγραφα ταυτότητα που θα αναγνωρίζουν τα άλλα κρατημέλη αν χαθεί, αν υπάρξει απώλεια. Για το διαβατήριο ισχύει ήδη, λέω πρέπει να ισχύει και για την ταυτότητα. Πρέπει απώλειες ταυτότητας να εκδίδεται ένα ε, έγγραφο που θα αντικαθιστά και θα το αναλάβουν οι προξενικές αρχές. Τελευταίο στοιχείο. Ίσως θα υπάρξουν αντιδράσεις. Θεωρώ ότι η ταυτότητα δεν είναι ένα σύμβολο εθνικής, εθνικού ανήκειν, ανήκειν σε μια χώρα, γιατί μπορεί κανείς με την ταυτότητα αυτή να κυκλοφορεί ελεύθερα στην επικράτεια της Εύρωσης και Ένωσης και το χρησιμοποιεί και για να εισέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα έχει ευρωπαϊκή διάσταση το έγγραφο αυτό. Και αυτό πρέπει να είναι σαφές. Ήδη γίνεται με, το διαβατήριο. Προτείνω λοιπόν στη μελλοντική ταυτότητα να μπαίνει σε τετράγωνο μπλε το σύμβολο της εθνικής ε, και γύρω-γύρω τα αστέρια της Ευρωπαϊκής Σημαίας. Τα έχω πει και στους Κιώδης, δύο φορές έχουμε συναντηθεί. Θα έχουμε την Τρίτη, την επόμενη εβδομάδα, πρωί Τρίτης, και άλλη μια συνάντηση και θα συνεργαστώ μαζί τους στενά στο βαθμό που θεωρώ ότι αυτό είναι σύμβατο με τους στόχους ε, του εγγράφου αυτού. Θα υπόψη, θα λάβω υπόψη τις στάσεις και τις κριτικές των συναδέλφων. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Ένας συνάδελφος μπορεί να μιλήσει, τουλάχιστον για ένα σκιώδη, για το ΕΛΚ. Μπάρμπαρα, μιλάς για τον Κάλλος Κοέλιο, για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Λέει ο Κάλλος Κοέλιο ότι δεν μπορούσε να είναι παρόν λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Δυστυχώς ήταν ανέφικτο να διεξαχθεί το πρωί η εξαγωγή της ε, συνεδρίας αυτής και μου ζήτησαν να σε διαβιβάσω μερικές σκέψεις του. Οι ταυτότητες, οι άδειε διαμονής είναι πολύ σημαντικά έγγραφα στον τομέα ελεύθερης μετακίνησης. Η πρόταση αυτή πετυχαίνει τρεις στόχους. Προωθεί την ελεύθερη μετακίνηση, καταπολεμεί την απάτη ταυτότητας και τέλος καταπολεμά την πλαστογράφηση των ταυτοτήτων σεβόμενος πάντα, σεβόμενη η πρόταση ε, το δικαίωμα των κρατών μελών έχει τις κάρτες. Ο κ. Ντεπρέ λοιπόν παρουσίασε την πρόταση, η έκθεσή του είναι καλή και γενικά μπορούμε να τη στηρίξουμε. Όμως, σαν σκιώδης εισηγητής ο κ. Κοέλιο θα ήθελε να τονίσει τέσσερα σημεία. Πρώτον, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι αυτή η πρόταση δεν καλύπτει το θέμα παραγωγής ε, των αρχικών εγγράφων, των εγγράφων που οδηγούν στην έκδοση ταυτότητας. Αυτά λοιπόν τα αρχικά τα έγγραφα, τα προαπαιτούμενα έγγραφα, ποικίλουν σε εθνικό επίπεδο ακόμα παραπάνω και καλύπτονται από λιγότερα μέτρα ασφαλεία. Δεύτερον, σε πλήρη σεβασμό της ε, γνωμοδοτήσεως περί υποστηρίζουμε ε, τη συλλογή βιομετρικών στοιχείων, αλλά δεν βλέπουμε γιατί παιδιά κάτω των 12 ετών δεν θα έπρεπε να δίνουν δαχτυλικά αποτυπώματα. Έχει αποδειχθεί από το κοινό κέντρο ότι τα δαχτυλικά αποτυπώματα ετών ε, παιδιών δημιουργούν λιγότερα προβλήματα από ότι ένα, ενός ατόμου 70 ετών. Για να έχουμε και άλλους τρόπους ταυτοποίησης, θα προστατεύουμε καλύτερα τα παιδιά σε περίπτωση διακίνησης ή απαγωγών. Οι ταυτότητες εκφράζουν εθνική ηθαγένεια, άρα και την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Δεν θέλουμε οι κάρτες της ταυτότητας να είναι οι ίδιες στην Ευρώπη. Όλοι. Θέλουμε οι ταυτότητες να τα αμοιβαία. Έτσι οι πολίτες να μην έχουν εμπόδια όσον αφορά την άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματος της ελεύθερης μετακίνησης. Τέταρτον, οι άδειε διαμονής πρέπει να δοθούν στα πλαίσια του, του συστήματος ενημέρωση ε, πληροφοριών Σέγγεν. Η υπήκοτή των χωρών, σύμφωνα με της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα μπουν στο σύστημα ΒΙΣ. Όποιο σύστημα συμφωνήσουμε, θα πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη. Προτιθέμε θα υποβάλουμε σχετικές τροπολογίες και προσβλέπουμε σε συνεργασία με τον εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητές. Και ελπίζουμε να εγκριθεί γρήγορα έκθεση. Το θεμελιώδη δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ενώσης είναι εξίσου σημαντικό όπως το δικαίωμα στην ασφάλεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μπάρμπαρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάτι να πει πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω είναι. Κύριε Μουζοβά. Ναι, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και που αποδίδετε τόση σημασία σε αυτήν την σημαντική πρόταση της Κομισιόν. Η πρόταση αυτή, όπως ήδη έχουν δηλώσει οι συγητές, αφορά την ελευθερία μετακίνησης των Ευρωπαίων πολιτών το να έχουν αξιόπιστα δελτία ταυτότητας, κάτι το οποίο βεβαίως ε, θα τους διευκολύνει. Η πρόταση, όπως αναφέρατε και εσείς ε, και οι σκιώδεις το στόχο έχει ακριβώς να κλείσει το κενό ασφαλείας. Τα δελτία ταυτότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διασχίσει κανείς τα εξωτερικά σύνορα, οπότε πρέπει να είναι πάρα πολύ ασφαλής. Γι' αυτό επιλέξαμε για μια πρόταση η οποία θα έχει και φωτογραφία και δακτυλικό αποτύπωμα γιατί αυτός ο συνδυασμός μπορεί να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε τις νέες τεχνικές απάτης και πλαστογραφίας. Σε γενικές γραμμές λοιπόν ευχαριστώ τον κύριο Ντεπρές για το σχέδιο έκθεσης. Πράγματι η πρόταση αυτή συμφωνεί με τους κύριους στόχους και τις αρχές της πρότασης και ελπίζουμε να μπορέσουμε να τον στηρίξουμε στις μελλοντικέ συζητήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ για την Προεδρία η κυρία Ταμάρα Κέρμπελ. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας πω λίγα λόγια για τη δουλειά που κάνει το Συμβούλιο. Η εξέταση της πρότασης ξεκίνησε στις 29 Μαΐου επί Βουλγαρικής Προεδρίας. Έκτοτε είχαμε τέσσερις ε, συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας. Έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος. Η πρώτη συνεδρίαση του σχετικού Συμβουλίου θα λάβει χώρα την επόμενη εβδομάδα και από εκεί θα συνεχίσουμε την δουλειά μας και ελπίζουμε να υπάρχει μια έντολη για διοργανικές διαπραγματεύσεις τον Νοέμβριο. Η Αυστριακή Προεδρία σας διαβεβαιεί ότι θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε μια συμφωνία στο Συμβούλιο και ότι αναμένουμε την συνεργασία μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιστρέφουμε λοιπόν στον Ζεράρ για τα τελικά του λόγια. Πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω καταρχάς τον κύριο Κοέλιο, τον οποίο αντικαθιστά πάνω από επάξια, για να πω κάτι άλλο, συνάδελφος, για το στοπιτικό παρουσίας. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Στην Πορτογαλία, αν έχω ακριβείς πληροφορίες, τα δακτυλικά αποτυπώματα τα παίρνουν από τη γέννηση. Για να εγγραφεί στο ληξιαρχείο το παιδί. Πώς? Όχι. Oui, oui. Bon, dès sont à ou en tout cas très... Α, όταν πάνε σχολείο. Τέλο πάντων όπως και αν έχει, πολύ νωρίτερα από τις άλλες χώρες. Και πρέπει να τα δούμε κατά πόσο είναι σκόπιμο. Να το δούμε στην έκθεση αυτό το θέμα. Για τα υπόλοιπα, σημειώνω τις προτάσεις του κύριου Κοέλιο και φυσικά θα τις εξετάσω. Με τη μέγιστη προσοχή. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την Κομισιόν που είπε ότι αν τη χρειαστούμε θα μας τίνει χείρα βοηθείας τα είπε πολύ ωραία και το Συμβούλιο επίσης, το ευχαριστώ που έδειξε προθυμία να συνεργαστούμε για να καταλήξουμε σε μια διοργανική συμφωνία το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστώ. Thank you very much, uh, Mr. Ευχαριστούμε κύριε Ντεπρέ. Μπάρμπαρα, συνάδελφοι. Α, ναι, προθεσμία κατάστροπολογιών. 9 Οκτωβρίου. 16 απόγευμα. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα στο 16. Στην ακρόασή μας. Είστε έτοιμοι όλοι για να δω. Um, Θα χαιρόμουν πολύ αν το πρώτο πάνελ ε, ομιλητών μπορεί να έρθει εδώ στο έδρανο. Θα ήταν υπέροχο κάτι τέτοιο. Και μετά θα ξεκινήσω κάνοντας την παρουσίαση. Θα του συστήσω. Um, Καλώς. Καλωσορίζω θερμά όλους τους ομιλητές. Καλωσορίζω θερμά όλους τους προσκεκλημένους που ήρθαν εδώ ειδικά για αυτή τη σημαντική ακρόαση που είναι και ευαίσθητη για την οδηγία διευκόλυνσης και για ανθρωπιστική βοήθεια στους παράτυπους μετανάστες όπως αποκαλούνται. Να πω καταρχάς κάτι εκφραζόμενος εκ μέρους των συναδέλφων. Είναι πολύ στεγνός, ξερός αυτός ο τίτλος. Αλλά το θέμα πρέπει να εξεταστεί ειλικρινά. Είναι μια από τις μεγάλες ε, τραγωδίες που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια ανθρώπινη τραγωδία είναι αυτή. Άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους. Τεράστια τραγωδία που συνεχίζεται τώρα που μιλάμε. Στη συζητήσεις σας σήμερα πρέπει να καταλάβουμε Ποια είναι η ανθρώπινη διάσταση. Δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Ποτέ. Αυτό που συζητούμε σήμερα στην ακρόση ακούγοντας τους συναθριστέντες εμπειρογνώμονες, είναι το θέμα της εφαρμογής της οδηγίας διευκόλυνσης, όπως αποκαλείται, στα κράτη-μέλη. Και πώς η ανθρωπιστική βοήθεια που χορηγεί τους μετανάστες και τους πρόσφυγες ε, δεν εφαρμόζεται σωστά. Είναι έγκλημα, τελικά τι γίνεται, είναι ένδειξη ανθρώπινης ε, αλληλεγγύης και πού βρίσκονται διαχωριστικές γραμμές. Γι' αυτό είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Το συζητήσαμε και όταν εκπονήσαμε ένα ψήφισμα πρόσφατα από την Επιτροπή μας προσήλκησε πολύ ενδιαφέρον. Αναφέρεται σε ένα τα μεγάλα διλήμματα. Πώς οι άνθρωποι, οι διάφορες οργανώσεις, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις μπορούν να σώσουν ζωές, αλλά δεν πρέπει να ποινικοποιούνται κατά την εκτέλεση αυτού του έργου. Περίπλοκη κατάσταση. Τα τελευταία χρόνια είδαμε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δικάζονται γιατί βοήθησαν ανθρώπους που αντιμέτωπιζαν προβλήματα και από την άλλη είπαμε διακινητές. Με τα μάτια μου το είδα αυτό. Έχοντας μεταβεί στη Λιβύη, στο εσωτερικό της Λιβύης, ότι οι διακινητές ωφελούνται από τους ευάλωτους ανθρώπους που παλεύουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να επανενωθούν με τις οικογένειές τους ή να τύχουν προστασίας ή να βρουν καλύτερο μέλλον. Δύσκολη ισορροπία. Το ξέρουμε πολύ καλά, κυρίως στην Επιτροπή μας. Απ' τη μία έχουμε την ανάγκη να τιμωρηθούν και να αποτραπούν οι διακινητές μέσω ποινικών κυρώσεων και απ' την άλλη πρέπει οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορούν να εκφράσουν ανθρώπινη αλληλεγγύη χωρίς να κινδυνεύουν με ποινικοποίηση. Ποινικοποίηση λοιπόν διακινητών από τη μια και απ' την άλλη έχουμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη μεγάλη από ανθρωπιστική βοήθεια. Καρπός της συζητήσεως είναι το πακέτο διευκόλυνσης. Συμπεριλαμβάνεται η οδηγία του 2002 και η απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου που εφαρμόζει την οδηγία. Με την πάω των ετών φάνηκε ότι η εφαρμογή του όλου πακέτου δημιούργησε νομική αβεβαιότητα και αμφισημία. Και πρόσφατα, όπως ανέφερα, το Κοινοβούλιο πρωτοβουλία αυτή τη Επιτροπής της ΛΥΜΠΕ κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκδώσει καθεδρίες γραμμέ προς τα κράτη-μέλη ώστε να αποφευθεί η ποινικοποίηση ανθρωπιστική βοήθειας μέσω του ψηφίσματο που ζητήθηκε 5 Ιουλίου. Βέβαια αυτό ακολούθησε την έκθεση Ματσόλα Κιέγγε, που συζητήθηκε εδώ, που ανέφερε και παραθέτει οποιοδήποτε παρέχει διαφορετικέ μορφέ ανθρωπιστική βοηθεία σε εκείνους που τη χρειάζονται, δεν θα πρέπει να ποινικοποιείται και θα πρέπει αυτό να αντικατοπτρίζεται σαν αρχή στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Και αυτή είναι η έκθεση που θετήθηκε και από την παρούσα Επιτροπή και από το Ευρωκοινοβούλιο. Χαίρομαι λοιπόν που καλωσορίζω του σημερινού φιλοξενούμενου μα. Θα μα βοηθήσουν να προχωρήσουμε περαιτέρω σε αυτό τον τομέα που είναι πολύ ενδιαφέρον αλλά και επίμαχο. Και θα ξεκαθαρίσουμε ποια είναι η γραμμή μεταξύ εκείνων που πραγματικά βοηθούν και εκείνων που κέρδο, βγάζουν κέρδος από την εκμετάλλευση αυτού. Να ακούσουμε συναδέλφους από δύο, μάλλον δύο πολίτες που συμμετέχουν στη Μεσόγειο, στην παροχή βοηθείας του μετανάστες. Ο κ. Νέστερ και ο κ. Αλντίν, με, μεταξύ ο κ. Ζων Κρούν, θα παρουσιάσει την άποψη των κρατών μελών και μετά θα στραφούμε προς τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ενώσης. Ο κ. Λετζέρη θα μιλήσει για τη Frontex, για το θέμα αυτό και τον κύριο Θοδωράκη από τη μονάδα υπεύθυνη για την καταπολέμηση της διακίνησης την DG Home της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα μέλη εδώ που έχουν εμπειρία στο θέμα και κάποιοι έχουν επισκεφτεί τις περιοχές αυτές και κάποιοι συνέβαλαν στο σημαντικό το, το ψήφισμα που πέρασε να εκφράσουν την άποψή τους. Ξεκινάμε. Πρώτο κομμάτι παρουσίαση προκατακτικών πορισμάτων. Από τη μελέτη Οδηγία Διευκόλυνσης ποινικοποίηση Ανθρωπιστικής Βοήθειας που παρέχεται προς τους παράτυπους μετανάστες. Θα ξεκινήσουμε αυτή την παρουσίαση. Η Λίζα Βασιλιούτα θα το παρουσιάσει, που συμμετέχει στο σχετικό πρόγραμμα στο ΣΕΠΣ και επίσης κάνει μεταδιδακτορικό στο Διεθνές Κέντρο Ανάπτυξη του Λονδίνου και στο κέντρο Σόλας, ΣΟΑΣ στο Λονδίνο για το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Μακροσκελέστατος τίτλο. Τα ξέρω τα μέρη που αναφέρω, δεν έπρεπε να μπορώ να τα αναφέρω. Η Λίνα και η Τζένιφερ λοιπόν. Αν μπορείτε να ξεκινήσετε παρουσιάζοντα τα προκατακτικά πορίσματα της μελέτης για την οδηγία διευκόλυνσης θα ήταν μια καλή αφετηρία. Έτσι θα έχουμε ένα πλαίσιο για την οδηγία. Λοιπόν, εναρκτήριο λάκτισμα. Αυτή η ακρόση μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Πέμπτη απόγευμα δεν έχουμε πολλά μέλη, ευχαριστώ τους παρόντες, αλλά μεταδίδεται στο διαδίκτυο ε, η εκδήλωση αυτή και παρακολουθούν πολλοί ακροατές και θεατές και δίνω το λόγο τώρα στους ε, καλεσμένους. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας και είναι μεγάλη μας χαρά που παρουσιάζουμε τα ευρήματά μας εδώ πέρα. Εκπροσωπούμε και άλλες συγγραφείς, ε, την κυρία Σάντσες και τον κύριο Καρέρα. Και η μελέτη αυτή βεβαίως βασίζεται και στην προηγούμενη έρευνά μας για τις πολιτικές ε, κατά της διακίνησης ε, και η διασταύρωση με την ανθρωπιστική βοήθεια που κάναμε το 16-17 όπως επίσης ε, και το τωρινό μας έργο όπου εστιάζουμε ιδιαίτερα στην καταστολή των ΜΚΟ και έχουμε και στο βάθος της αίθουσας υλικό για όσους ενδιαφέρονται. η μελέτη η ίδια θα οριστικοποιηθεί στα τέλη Οκτωβρίου αλλά δεν είναι άρα δημόσια αλλά ελπίζουμε να βοηθήσει στο ψήφισμά σας και στις περαιτέρω προτάσεις σας για το πώς μπορεί να εξαιρεθεί η ανθρωπιστική βοήθεια. Επίσης, ε, έχουμε κάνει μια έποψη ε, της παρακολούθησης των ΜΜΟ που παρακολουθήσαμε ακριβώς την εκτεταμένη ποινικοποίηση της αλληλεγγύης και της ανθρωπιστικής βοήθειας ε, και αυτοί οι οποίοι ποινικοποιούνται είναι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και δημοσιογράφοι, πάροχοι υπηρεσιών και επαγγελματίες όπως οι δικηγόροι. Οπότε το εύρος ε, είναι μεγάλο και πηγαίνει πέρα από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις και όταν βλέπουμε τις συνθήκες που οδήγησαν ε, στην κατάσταση αυτή της ποινικοποίηση βλέπουμε ότι η ασάφεια του εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου είναι ένα βασικό ζήτημα εδώ. Δεύτερον, έχουμε την επίγουσα φύση της κατάστασης της καταπολέμησης ε, της διακίνησης ε, και έτσι το ποινικό δίκαιο υπάγεται στην ε, καταπολέμηση της διακίνησης οπότε δεν είναι σαφές το τι κάνουν οι αστυνομικοί όταν, τη στιγμή που συλλαμβάνουν κάποιον. Και υπό το φως αυτής λεγόμενης ε, κρίσης ε, είχαμε κυρίως μονομερείς αντιδράσεις και όχι ευρωπαϊκές. Οπότε βλέπουμε ο καθένας να κοιτάει το συμφέρον του, το κάθε κράτος μέλος, να μετατοπίζει την ευθύνη σε άλλα κράτη-μέλη ή στην κοινωνία των πολιτών, όπως παραδείγματο χάρη στην κατάσταση της έρευνας και διάσωσης και το ποιος είναι υπεύθυνο. Επόμενο. Οπότε, όπως, ως ένα πρώτο στοιχείο, το κείμενο της οδηγίας ε, λέει ότι οποιαδήποτε εσκεμμένη βοήθεια για είσοδο ή διέλευση ανεξαρτήτως ε, πρόθεσης ποινικοποιείται οπότε σύμφωνα με την ανάλυση μας και ως αυτό ευθυγραμμίζεται και με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές ε, περί υλικού ωφέλους δεν υπάρχει ε, το ποινικό στοιχείο ή πρόθεση γιατί ε, θεωρούνται εγκληματικές αυτές οι πράξεις. Επόμενο. Όπως βλέπουμε αυτήν την στιγμή μόνο 4 από τα 26 κράτη-μέλη έχουν ευθυγραμμιστεί με τις προδιαγραφές του ΟΗΕ, δηλαδή να ζητάνε ουσιαστικά ή άλλα οικονομικά ωφέλη για να διώξουν ε, την ε, διακίνηση, δηλαδή η Γερμανία, η Ιρλανδία, Λουξεμβούργο και η Πορτογαλία. Τα υπόλοιπα κράτη-μέλη ακολουθούν την παρέκκληση του σχετικού πρωτοκόλου του ΟΗΕ που βασικά λέει ότι οποιαδήποτε υψηλότερη ε, ποινή ισχύει. Όμως ε, με αυτόν τον τρόπο αντιβαίνουν στον στόχο του πρωτοκόλου παράνομης διακίνησης του ΟΗΕ. Όταν μιλάμε τώρα για τους ε, κατοίκους, ε, ο νόμος απαιτεί να υπάρχει οικονομικό όφελος, όμως ακόμα τα μισά κράτη-μέλη δεν είναι πεπισμένα ότι θα πρέπει να απαιτούν ε, να υπάρχει το στοιχείο αυτό για να ασκήσουν διώξεις. Επόμενο και εδώ πέρα το σημαντικότερο, σημαντικότερη διάταξη που αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξαίρεση ανθρωπιστικών δράσεων. Η τωρινή οδηγία το αφήνει στα χέρια των κρατών μελών να αποφασίσουν εάν θα ποινικοποιήσουν ή όχι την ανθρωπιστική βοήθεια ε, εν τη της. Επόμενο. Και πάλι αυτό δεν ευθυγραμμίζεται με τις προθέσεις ε, του σχετικού πρωτοκόλλου του ΟΗΕ όπου λένε ότι ο λόγος για τον οποίο απαιτείται να υπάρχει κέρδος είναι ότι είναι ακριβώς να μην τιμωρηθούν ομάδες οι οποίες το κάνουν για λόγους ανθρωπιστικούς ή αλτροιστικούς, όπως γίνεται στην περίπτωση έτουν άσυλο. Και έχουμε κάποιες μορφές ρητών εξαιρέσεων σε Βέλγιο, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Μάλτα και Ηνωμένο Βασίλειο. Όμως σε κάποιες από αυτές τις χώρες είχαμε πάλι διώξεις ε, και σήμερα θα ακούσουμε μια τέτοια περίπτωση από δύο χώρες όπου συνεχίζονται οι διώξεις. Επόμενο. Και καμιά φορά ακούμε ότι δεν είναι σαφές το ότι πρέπει να εξαιρεθεί όμως όταν κοιτάμε το ευρωπαϊκό κονσένσους, την συνένεση ε, φαίνεται ότι ο στόχος είναι σαφής. Έχουν συμφωνήσει τα κράτη-μέλη και λέει ο στόχος να διασωθεί η ζωή, να μην, να μην υποφέρει κάποιος, ε, να προστατευτεί η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, εάν ε, το κράτος ή οι τοπικοί φορείς δεν θέλουν ή δεν μπορούν να δράσουν. Και αν δούμε την έρευνα και η διάσωση, η συνένεση αυτή, η συνεννόηση θα μπορούσε να εφαρμοστεί ευρέως. Και αν την εφαρμόζουμε για τρίτες χώρες, γιατί να μην εφαρμοστεί και εντός της Ένωσης. Επόμενο. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα ζητήματα όπως η νομική αμεβαιότητα μεταξύ των παρόχων της υπηρεσίας ε, με το τωρινό πλαίσιο της Ένωσης υπάρχει ε, διαφορετική εφαρμογή στα κράτη-μέλη και ποινικοποίηση των μεταναστών που είναι θύματα της διακίνησης. Και υπάρχουν δυσανάλογες ποινές. Επόμενο. Λοιπόν, θα αναλάβω εγώ. Όπως είπε και η Λίνα, η έρευνα αυτή βασίζεται σε έργο το οποίο είχατε αναθέσει ως Επιτροπή ε, σε μας, αλλά και σε μια μελέτη από το, που τη χρηματοδότησε το Οικονομικό Ερευνητικό Συμβούλιο για Ουγγαρία, Ιταλία, Ελλάδα ε, και την Ένωση συνολικά βέβαια, κυρίως όμως στις χώρες αυτές. Και κάτι το οποίο προέκυψε είναι ότι δεν μιλάμε μόνο για την ποινικοποίηση, για τη δυναμική επίσης ε, της ποινικοποίηση ΜΚΟ και οργανώσεων της κοινωνίας ε, των πολιτών ε, μέσω και μέχρι και διώξεων. Δεν θα χρειαστεί βέβαια κανείς να φυλακεί στα σίδερα για να βιώσει τι θα πει ποινικοποίηση. Είδαμε λοιπόν τέσσερα βασικά στοιχεία στα κράτη-μέλη διαφορετικές μορφές, ε, υποψία και καχυποψία, μέτρα πειθαρχικά, εκφοβισμός, παρενόχληση και τέλος η δίωξη. Αυτή καθεαυτή. Δεν θα μιλήσω για τη δίωξη, γιατί και η Λίνα είπε ότι υπάρχουν συνάδελφοι που θα σας ε, μεταφέρουν αργότερα άμεσα τις δικές τους εμπειρίες. Το που εγώ θέλω να τονίσω όμως ε, σε σχέση με την ε, αστυνόμευση και τη διεξήνω. Αυτά που μας είπαν εθελοντές από οργανώσεις ε, της κοινωνίας των πολιτών, παραδείγματος χάρη στο Καλέ, ότι αυτό που βιώσανε ήταν ότι δεν τους προστάτευε η αστυνομία, ένιωθαν ευάλωτοι. Όταν δηλαδή έδιναν τρόφιμα στους ετούντες άσυλο, δεν τους προστάτευε η αστυνομία από τους διακινητές. Δηλαδή, πολλές φορές η αστυνομία ε, είναι ε, αντί να, τους ε, ε, δίνει κάποια μαθήματα ενδεχομένω είναι σαν να τους διώκει αυτούς. Άλλα παραδείγματα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ουγγαρία, ΜΚΟ έπρεπε να ε, τηρούν αυστηρούς κανόνες, ε, μέτρα, να είχαν πρόσβαση κάποιες μικιό σε κάποια κέντρα κράτησης στην Ουγγαρία συνέβη αυτό, καχυποψία, αυτό επιδεινώνεται από τα μέσα ενημέρωσης. Οι γιατροί χωρί σύνορα, για παράδειγμα, που είχαν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στα θαλάσσια και στα χερσαία σύνορα, υποστηρίζοντα ε, τους πρόσφυγες στη διάρκεια της κρίσης, τους κατηγορούσαν ε, ότι είναι σαν θαλάσσια ταξί και για τον εκφοβισμό και την παρενόχληση. Μπορείτε να διαβάσετε και το βιβλίο ή το έγγραφα που έχουμε αφήσει πίσω στην αίθουσα για να δείτε απειλέ, μέσα κοινωνική δικαιοσύνη, σωματικέ απειλέ, ε, παρενόχληση, να του ζητάνε για να δείξουν έγγραφα. Μέχρι και σεξουαλική κακοποίηση από την αστυνομία ή από τι ε, ε, μονάδε επιβολή του νόμου και σε βάρο ακτιβιστών χωρίς καν να τους επιδεικνύουν ταυτότητα, άρα δεν μπορούν να ερευνηθούν αυτά τα περιστατικά σωστά. Αυτά είναι λίγα από τα παραδείγματα, αλλά μπορείτε να βρείτε στη μελέτη μας πολύ περισσότερες πληροφορίες. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε λίγο πολύ γιατί μιλάμε εδώ. Μπορεί να είναι σχετικά μικρός ο αριθμός, πώς να το πω, ανθρώπων οι οποίοι σαπίζουν ε, στις φυλακές ε, για ε, αδικήματα. άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι επειδή προσπάθησαν να βοηθήσουν όπως ο κ. Λόρι που τον συνέλαβαν γιατί η πτάχα διακινούσε ένα παιδί που ήθελε να ε, βρει την οικογένειά του ε, στο Καλέ. Πάρα πολύ ε, αγχώδης εμπειρία, ευτυχώς αθώθηκε. Τι άλλο βλέπουμε. Δεν μιλάμε μόνο για τα δικαιώματα των μεταναστών αν και είναι ουσιαστικά αυτό το θέμα ε, και η ανθρώπινη ζωή, αλλά είναι και θέμα που έχει να κάνει τους πολίτες. Αυτό μας το λένε συνέχεια οι ΜΚΟ, αλλά και οι μετανάστες με τους οποίους μιλάμε και μιλήσαμε στο πλαίσιο της έρευνας. Τι κάνει η κοινωνία των πολιτών ουσιαστικά, προασπίζεται το δικαίωμά της να προστατεύει τους έχοντες ανάγκη. Είναι μια θεμελιώδης αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Γαλλία έχουμε τον κύριο Χεγό, ο οποίος πρόσφατα, πρόσφατα συνελήφθη ότι διακινεί ε, ανθρώπους από την Ιταλία στη Γαλλία. Ξεκίνησε μια συζήτηση στην ε, δίκη του τι θα πει αδελφότητα, αδελφοσύνη. Είπε ότι αυτό είναι, αυτό που κάνω εγώ. Θέλω να προστατεύσω τους αδελφούς μου. Θέλω να ενωθούν τις οικογένειες. Αυτό που έλεγε και ο Κλοντ. Τι θα πει να είναι κανείς Ευρωπαίος και να αγωνιστεί για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εδώ βλέπετε τις 170 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών άνευ προηγουμένου εκλίμακ. Μεγάλη ε, επίδειξη αλληλεγγύης. Αλλά με αφορμή την ε, λεγόμενη μεταναστευτική προσφυγική κρίση είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τόσο μεγάλη κινητοποίηση και αλληλεγγύη. Και εδώ κάποια παραδείγματα από πρωτοβουλίες που φαντάζομαι γνωρίζετε για να τεθεί υπόψη του Κοινοβουλίου το ζήτημα και χαιρόμαστε που έγινε αυτό γιατί πραγματικά ε, υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία, πάρα πολλές πληροφορίες ε, για όλους. Είναι πρώτη φορά που η Παγκόσμια Οργάνωση κατά των Βασανιστήριων άρχισε να παρακολουθεί το θέμα των προσπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρχίζει δηλαδή να προσελκύει το διεθνέ ενδιαφέρον. υπάρχει ε, υπάρχει δικαίωση συγητή ε, από τον ΟΗΕ για τα θέματα που παρακολουθεί. Πλέον υπάρχει μια δυναμική λοιπόν σε ό,τι αφορά όλες αυτές τις τέσσερις ε, κακές δυναμικές που είδα, που σας είπα, εκφοβισμό και Ε, και τα λοιπά, δημιουργούν ε, στιγματοποίηση, δημιουργούν προβλήματα αλλά ευαισθητοποιούνται και πολύ. Τι διακυβεύεται, δεν είναι μόνο η διάσωση ζώων στη θάλασσα, αλλά και στα χερσαία σύνορα. Είπαμε, διακυβεύονται τα δικαιώματά μα, τα δικαιώματα των Ευρωπολιτών, να μπορέσουμε να δώσουμε ένα κομμάτι ψωμί σε έναν που πεινάει και να μα κατηγορήσει κανεί. με βάση την ε, παραποίηση κάποιου διάταξη μιας ε, ενός νόμου και να καταδικάσετε κάποιος, να κατηγορείτε για διακίνηση, να πάει να βοηθήσει. Γίνεται συχνά λόγος για μείωση του αριθμού των ε, αφήξεων ε, των ε, νομότυπων μεταναστών. Η πραγματικότητα είναι ότι μπορεί μάλλον παράτυπων μεταναστών Ναι, έχει μειωθεί ο άνθρωπο των παράτυπων μεταναστών, αλλά έχει αυξηθεί ο άνθρωπο αυτών που πέθαναν στην προσπάθειά του ε, να φτάσουν. Και που είναι και θέματα διακίνησης. Και είναι ανάλογη αύξηση ε, της αύξησης και της αστυνόμευσης και των ε, προσπαθειών ε, που κάνουν οι αρχές από το φυλακή Είναι τροφή για σκέψη αυτό. Κάτι πιο γενικό. Πώς μας επηρεάζουν όλα αυτά. Από την έρευνα, την παρελθούσα γνωρίζουμε ότι τα μέτρα τι αποτέλεσμα έχουν. Αποτροπή ε, για τις φιλανθρωπικές οργανώσεις που δεν εργανώνονται πια τόσο για να βοηθήσουν. Στο Ρωμένο Βασίλειο οι νοικοκύριδες, οι διοκτήτες ε, ζητάνε από τους ε, ενοικιαστές τους ε, πάρα πολλά έγγραφα που να πιστοποιούν την καταγωγή τους. Και αν το όνομα κάποιου ακούγεται ξένο, πολλές φορές δεν θέλουν να νοικιάσουν το σπίτι τους. Και επίσης αυτά ανοίγουν την πύλη και για την κατάργηση του κράτους δικαίου. Δεν προωθούνται οι αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης. το δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση για τα συνολικά παιδιά. Δε, πολλά χρόνια χρειάστηκε για να αρχίσει να αλλάζει κατάσταση και να κινούνται τα πράγματα και αυτό χάρη στη ΜΚΟ. Και επίσης χρειάζεται και περισσότερη ασφάλεια, ε, συγγνώμη, σαφήνεια δικαίου. that it uh, has... Κοιτάξτε, Υπάρχουν και δυνατότητες να διευκαθούν και άλλες μορφές εγκλήματος που έχουν ε, διαπράττονται πραγματική εγκληματική πρόθεση και είναι αντικείμενο διακίνησης και εκμετάλλευσης οι πρόσφυγες. Κάποιες συστάσεις. Συμφωνώ με τη θέση του Κοινοβουλίου. Πρέπει να καθορίσουμε τη διαχωριστική γραμμή τι ποινικοποιείται και τι δεν ποινικοποιείται. Είδαμε το προηγούμενο στην Οδηγία της Ευρωπαϊκής για την διακίνηση ανθρώπων που εξαιρεί τα θύματα της διακίνησης. Παρομοίως, εκείνοι που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια θα μπορούσαν να εξαιρεθούν από την ποινικοποίηση. Επόμενο. Όπως είδαμε, παρά το ότι κάποια κάτι μέλη έχουν σωματώσει νομοθεσία του την ανθρωπιστική εξαίρεση, στην πράξη δεν εφαρμόζεται. Πρέπει να υπάρξουν εποπτικοί μηχανισμοί που θα λειτουργούν. Το ελεκτικό συνέδριο, Φερρυπίν. Να παρακολουθεί κατά πώς χρησιμοποιούνται τα χρήματα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεως και κατά πόσο η καταπολέμηση της διακίνησης των ανθρώπων, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται συνάδει με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και Ευρωπαίος συνήγος του πολίτη θα πρέπει να εξετάζει και τι αξιολογήσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αν δούμε να αυξάνεται ο ρυθμό θανάτων στη Μεσόγειο, κάτι θα πρέπει να πηγαίνει στραβά με τι τρέχουσε πολιτικέ. Τρίτον, ανεξάρτητο παρατηρητήριο που δημιουργείται μαζί με πανεπιστημιακού ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και κοινωνία των πολιτών. Θα μπορεί να καταγγέλλεται τι υποθέσει κοινωνία των πολιτών και θα πρέπει να συνδέεται αυτό με την χρήση της νομοθεσίας και να εντοπίζεται αν υπάρχει σοβαρή συστηματική ε, παράβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή αν δίνεται μια πολιτική χρειά στις πράξεις. Τρίτον, συμφωνούμε με τη θέση του Ευρωκοινοβουλίου. Για να λυθεί το θέμα, πρέπει να ακολουθεί μια σφαιρική ολιστική προσέγγιση στη μετανάστευση. Μέχρι τώρα, μονόπλευρη περιοριστική πολιτική εφαρμόζεται, πολιτικές. Όταν εξετάσουμε εις βάθος το θέμα της διακίνησης μεταναστών, όταν υπάρχουν λιγότερες νόμιμες διέξοδοι για τους οικονομικούς μετανάστες και για τους πρόσφυγες και η δυνατότητα να έρθουν νόμιμα στην Ευρώπη χρησιμοποιούν τους διακινητές, αν δεν υπάρχουν αυτά δεν τροφοδοτούμε ε, το έργο των διακινητών και η έρευνα και διάσωση, οι πρακτικές αυτές είναι κάτι αναπόφευκτο σε, στην περίπτωση μονοπρευρών λύσεων. Και βλέπουμε τα κράτη που σπρώχνουν ένα στο, τη βάρκα στον άλλον όταν υπάρχουν βάρκες με πρόσφυγες. Σας ευχαριστώ. Να πω στους συναδέλφους ότι αυτό είναι το αρχικό έγγραφο που ζητήσαμε το 2016 και κάποιες από τις παρουσιάσεις ε, που ακούσατε προετοιμάζονται και για μια ενημέρωση του 2018 όπου θα έχουμε πιο ε, επίκαιρες πληροφορίες λοιπόν αυτά τα οποία συμβαίνουν ε, στην Μεσόγειο από αυτά τα οποία ε, μας είπατε νομίζω περιγράφουν την κατάσταση Αυτά λοιπόν για να σωστά παρακολουθείτε αυτά, περνάμε τώρα στον κύριο Νέστλερ, ιατρό και εθελοντή για διάφορες αποστολές ε, στην οργάνωση Lifeline Ships. Έχετε τον λόγο για 10 λεπτά. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω και να εκπροσωπήσω να εκπροσωπήσω κάποιες ε, οργανώσεις λέγομαι Nestler, ε, εργάζομαι στην αναισθησία και στη... επίγοντα στο Βερολίνο ε, πρώτα ξεκίνησα να εργάζομαι με τους μετανάστες και πρόσφυγες στο Βερολίνο, μετά στην Ελλάδα και μετά στην Κεντρική Μεσόγειο και ε, με πληρώνουν διάφορες γερμανικές ΜΚΟ για διάφορες αποστολές ε, σε διάφορα πλοία Juventa, Lifeline ε, και τα λοιπά. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρουσιάσω λίγο την περίπτωση της ε, κατάσχεσης των πλοίων Juventa και Lightline και της ποινική δίωξης ε, των μελών του πληρώματος. 2017 Juventa ξεκίνησε το 2015 και τον Αύγουστο του 2018 κατασχέθηκε Εν τω μεταξύ είχαμε διασώσει 14.000 άτομα που έφυγαν από τη Λιβύη. Όπως όλα τα πλοία στην περιοχή, η Γιουβέντα ήταν υπό τις οδηγίες του Ιταλικού Κέντρου Συντονισμού στη Ρώμη. Σώζαμε κόσμο από τον πνίγμο και βρίσκαμε και πάρα πολλά πτώματα, τα οποία επίσης φέρναμε στην Ιταλία. Στις περισσότερες περιπτώσεις ε, τους παραδίδαμε σε σκάφη της ακτοφυλακής του ΝΑΤΟ. Στις περιπτώσεις αυτές ακολουθούσαμε το εθνικό και διεθνές δίκαιο και συνεργαζόμασταν πλήρως με όλες τις αρμόδιες αρχές. Στις αρχές ε, του 2017 οι Ιταλικές αρχές άρχισαν να μας ερευνούν. Πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών και η αστυνομία καταπολέμησης της μαφίας ε, ε, είχε στόχο να μπει στο πλήρωμα των πλοίων, να παρακολουθεί τα τηλέφωνα και να βάλει και κοριούς στη γέφυρα του πλοίου. Για να γίνουν αυτά, πολλές φορές η Γιουβέντα διατάχθηκε να φύγει από την ζώνη ανοιχτά της Λιβύης και να κατευθυνθεί στο λιμάνι της ε, Λαμπεδούζας. Και εγκαταλείψαμε σε αυτές τις περιπτώσεις διάφορες βάρκες και δεν ξέρουμε τι απέγιναν. Ε, κάποιες από αυτές χάθηκαν τελικά τον Αύγουστο του 2018 η Γιουβέντα δεσμεύτηκε στο λιμάνι της Λαμπεντούζα κατόπιν εντολής ε, του Ισαγγελέως και κατηγορηθήκαμε για διευκόλυνση παράνομης ε, μετανάστευσης 22 ε, άτομα, 10 ήταν μέλος του πληρώματος. Ήδη οι εισαγγελείς αναγνώρισαν ότι δεν έχει υπάρξει κάποιο οικονομικό όφελος των ΜΚΟ, ούτε είχαν σχέσεις με λαθροδιακίνητες. Όμως οι αρχές έλεγαν ότι το Γιουβέντα ήταν μέρος μιας αλυσίδα που οδήγησε στην παράνομη είσοδο στην Ιταλική επικράτεια και άρα μπορεί να κατεργηθεί σύμφωνα με τον νόμο. Μετά την δέσμευση του Γιουβέντα, πολλές άλλες ε, ΜΚΟ ε, αντιμετώπισαν μια τεράστια καμπάνια με νομικά και γραφειοκρατικά εμπόδια για να μην συνεχίσουν να σώσουν ζωές. Τον Ιούνιο του 2018 το πλοίο Lifeline δεν μπορούσε να δέσει σε ευρωπαϊκά λιμάνια αφού διέσωσε 234 άτομα. Η λεγόμενη Λιβυιακή ακτοφυλακή ζήτησε να τις παραδοθούν οι μετανάστες για να επανέλθουν στη Λιβύη. Ο πλοίαρχος, ο Κλάς Ράις, ε, αρνήθηκε να υπακούσει στην διαταγή και επέμενε ότι θα έπρεπε να πάνε σε ένα λιμάνι όπου δεν θα υπήρχε η απειλή εκβιασμού ή βιασμού. Κατόπιν τούτου η Ιταλία και η Μάλτα ε, αρνήθηκαν να δώσουν ε, κάποιο λιμάνι στο οποίο θα μπορούσε να δέσει το πλοίο. Το πλοίο αναγκάστηκε να μείνει στα ανοιχτά για έξι μέρες ε, με πολλούς άρρωστους και ανήλικους. Τελικά του επιτράπη να δέσει στην ε, Μάλτα αφού ε, υπήρξε μια συμφωνία με πολλές κυβερνήσεις για να δεχτούν τα άτομα. Όμως κατόπιν οι αρχές της Μάλτας κατηγόρησαν τον κυβερνήτη για διαφορές παρανομίες που αφορούσαν το νεολόγιο του πλοίου και τώρα ο κυβερνήτης αντιμετωπίζει φυλάξη ενός ε, χρόνου για παραβάση του νεολογίου παρά το ότι είχε Ολλανδική σημαία και έχει όλα τα σχετικά έγγραφα. Και αυτά τα έχει επιδείξει και στο δικαστήριο και δημοσίως. Ένα άλλο πλοίο διάσωσης, το Sea 3, έκτοτε δεν του έχει επιτραπεί να φύγει από το λιμάνι της Μάλτας χωρίς καμία εξήγηση. Το Aquarius, ε, το οποίο ε, λειτουργεί η, λειτουργούν οι γιατροί χωρίς σύνορα, θα χάσει προσεχώς την σημαία του, καθώς η Ιταλία παρενέβη στο Παναμέζικο νιολόγιο Και οι αρχές του Παναμά λένε ότι το Aquarius δεν είχε επιστρέψει τα άτομα στην Λιβύη, κάτι το οποίο παραβιάζει την ε, συνθήκη της Γενέβης, οπότε κανείς δεν έχει κάνει ούτε ε, πλοία ΜΚΟ ούτε η Frontex. Ως ε, μισό αποτέλεσμα αυτών των ε, δράσεων το ποσοστό θανάτου πλέον ανεβαίνει σε, ανέβηκε ένα άτομα στα 16, τέσσερις φορές παραπάνω από το ποσοστό στους πρώτους μήνες του έτους που ήταν ένα στους 64. Εάν κριθεί ένοχο το πλοίο του Ιουβέντα, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 20 ετών και πρόστιμα 20.000 ευρώ για κάθε άτομο που μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη βοήθειά τους. Είμαστε πεπισμένοι ότι τελικά θα αθωθούν, αλλά όπως έχουμε μάθει και από προηγούμενες περιπτώσεις, η διαδικασία αυτή μπορεί να τα βήξει πολλά χρόνια και να κοστίσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε νομικά έξοδα. Οι άνθρωποι οι οποίοι ερευνώνται τώρα είναι επαγγελματίες ναυτικοί, πυροσβέστες, διασώστες, πολιτισμικοί διαμεσολαβητές και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι άφησαν την ησυχία τους για να σταματήσει ε, ο θάνατος στην πόρτα της Ευρώπης. Δούλεψαν εθελοντικά για χρόνια. Έχω συναντήσει μεταξύ αυτών ε, τα πιο ευγενικά άτομα που έχω γνωρίσει ποτέ. Και τώρα να βλέπω να τους κατηγορούν ως εξτρεμιστές και εγκληματίες, να δικάζονται και να κινδυνεύουν με φυλάκιση πραγματικά με θλίβη και πραγματικά σοκαρίστηκα που γίνονται αυτά τα πράγματα σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντί να τιμούμε αυτούς τους ανθρώπους, ε, τους θεωρούμε εγκληματίες και τους σταματούμε και καταστρέφουμε τις ζωές τους. Ως ιατρός έχω την νομική υποχρέωση να βοηθήσω σε οποιαδήποτε κατάσταση ανάγκης. Χωρίς καμία διάκριση δεν μπορεί να είναι η ευθύνη των ιατρών και των λοιπόν να αξιολογήσουν τη νομική κατάσταση ατόμων πριν δώσουν βοήθεια. Φοβούμε ότι εάν συνεχίσει έτσι η δίωξη ανθρωπιστών για πολιτικούς ε, στόχους θα υπονομευτεί η θέληση ατόμων να βοηθήσουν άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα σύνορά της. Γι' αυτό σας ζητώ να διαμορφώσετε ένα δεσμευτικό νομικό πλαίσιο που θα προστατεύει τον ανθρωπισμό από τις διώξεις που βλέπουμε σήμερα που ε, θα διακρίνει ξεκάθαρα μεταξύ αυτών που κερδίζουν από αυτή την υπόθεση και αυτών που δεν κερδίζουν. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δόκτωρα Χέσλερ. Προχωράμε. Ακούσουμε άλλο συνάδελφο που είναι στην πρώτη γραμμή. Σάρα Μαλτίν, την Team Humanity, τη και ΜΚΟ δημιούργησε, που κατηγορήθηκε για διακίνηση στη Λέσβο το, το 2018. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ που με καλέσατε και μου δείτε δυνατότητα να μιλήσω. Σαλάμ Αλντίν το όνομά μου. Θα θυμόσαστε τον Χόρντινγκ. πριν από τρία χρόνια. Το άψυχο σώμα του βρέθηκε στι τερκικέ αχθέ. Ήταν πρόσφυγα σύρος τριών ετών προσπαθούσε να θυτάσει ασφαλώ στην Ελλάδα. Είδα αυτή τη φωτογραφία που άλλαξε τη ζωή μου. Είδα τη φωτογραφία τότε στα νέα, ήταν τις 3 Σεπτεμβρίου του 2015. Τότε Ήμουν ένας απλός άνθρωπος, είχα μια δουλειά, ένα σπίτι, μια οικογένεια και φίλους. Τι περισσότερο μπορούσε να ζητήσει κανείς. Η εικόνα του Αιλάν Κουρντ ήταν, είχε κολλήσει στο μυαλό μου για μέρε και αναρωτιόμουν πώ μπορούσε ο κόσμο να το αφήσει αυτό, να το ξεχάσει το θάνατό του. Ο θάνατο αναθώου παιδιού που είχε μια οικογένεια που δεν θα του δώσει τίποτα περισσότερο από μια ευκαιρία για καλύτερη ζωή από, αντί να ζήσει σε μια εμπόλεμη χώρα και να μεγαλώσει εκεί. Και εγώ έχω προσφυγικό υπόβαθρο και μπορούσα να καταλάβω τον Αϊλάν. Είχα γεννηθεί στη Μολδαβία από Ιρακινό πατέρα και Μολδαβή μητέρα. Όταν ήμουν εννέα, έπρεπε να φύγουμε από τη Μολδαβία λόγω του εμφυλίου πολέμου. Ήταν μακρύ και σκληρό το ταξίδι, Περάσαν πολλέ χώρε πριν να φτάσουμε τελικά στην προορισμό μα που ήταν η Δανία. Εκεί μα αναγνωρίστηκε το καθεστώ των προσφύγων. Η φωτογραφία του ε, του Άλαν τσίγκλισε την συνείδησή μου και έγινε μια κλίση για δράση. Δεν μπορούσα να καθίσω εκεί με σταυρωμένα τα χέρια. Αν συνεχίσουμε να γνωρούμε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, θα πρέπει να δούμε ότι το, το αίμα έχει ε, λεκιάσει τα χέρια μας. Έπρεπε να κάνω κάτι. Λοιπόν, δύο μέρες μετά από τη φωτογραφία στα γενέθλιά μου στις 5 Σεπτεμβρίου αποφάσισα να πετάξω στην Ελλάδα για μια εβδομάδα να βοηθήσω. Τρεις ώρες μετά που προσγειώθηκα στο αεροδρόμιο της Λέσβου ήδη κολυμπούσα προς τα σκάφη ε, των, των προσφύγων που είχαν κολλήσει μερικά σε εκατοντάδες μέτρα από την ακτή και βοηθούσαν να σωθούν άντρες, γυναίκες, παιδιά και μικρά νεγέντα παιδιά. Δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε και είχα συγκλονιστεί. Δεν έβλεπα μεγάλες οργανώσεις, μόνο ΜΚΟ που έδιναν νερό και μπανάνες. Πού ήταν η ελληνική κυβέρνηση, πού ήταν ο ΙΕ, πού ήταν ο Ιθρός Σταυρός, πού είναι η αστυνομία. Αυτή η εβδομάδα μου άλλαξε εντελώ τη ζωή. Δεν κοιμήθηκα όλη την εβδομάδα. Επέστρεψα στη Δανία, μίλησα με φίλου και τρει μέρε αργότερα, με περίπου 30 ανθρώπου σε τρία πουλμανάκια, πήγαμε στη Λέσβο για την ανθρωπότητα. Έτσι ιδρύσαμε τη ΜΚΟ μα. Και έτσι ξεκίνησε η προσπάθειά μα να σώσουμε ζωέ. Ζωή, σταματήσαμε τη ζωή μα, ούτω ώστε να σώσουμε τη ζωή των προσφύγων. Άοκνα εργαζόμαστε 24 ώρες 24 ώρο, ε, περιπολώντας την αχτή μέρα και νύχτα, ελπίζοντας να σώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ζωές. Μερικοί από εσά ίσως να πρέπει να σκεφτείτε γιατί είχαν ανάγκη αυτοί οι άνθρωποι. Ήταν παγωμένε θερμοκρασίε, ρεύματα και οι γυναίκε άντρε και παιδιά και ηλικιωμένοι ήταν στριμωγμένοι σε μικρά ε, φουσκωτά σκάφη που ήταν πολύ μικρά και πολύ ασταθή για ανοιχτή θάλασσα. Αυτά δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν σε τόσε μεγάλε αποστάσει στη θάλασσα. Παρ' όλα αυτά επεμείναμε στη δουλειά που κάναμε, σώζοντας καθημερινά ζωές, όσο μπορούσαμε δηλαδή. Καμιά φορά αυτό δεν αρκούσε. Εγώ κρατούσα ανθρώπους που ξεψυχούσαν, που ξεψύχησαν στα χέρια μου και τα κορμιά τους πάγωναν. Αθώα παιδιά, αθώα βρέφη και πολύ συχνά ε, θυμάμαι τα τελευταία λόγια που μου είπαν θα πεθάνω ή βοηθήστε με. η όταν με ρωτούσαν οι οικογένειες αν θα επιβιώσουν οι αγαπημένοι τους. Εγώ ξέχασα πόσα παιδιά πέθαναν στη θάλασσα και εκείνα τα, τα, σώματα που ξεβράστηκα. Ε, ώρα περάσαμε ε, σκάβοντας τάφους για να θάψουμε ε, σώματα που δεν είχαν επιβιώσει από το ταξίδι για να φτάσουν στη Λέσβο. Ε, δεν ήρθα γι' αυτό εδώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι συνεχιζόμενα τα προγράμματα αυτά, τα προβλήματα, συγγνώμη, στον ανθρωπιστικό τομέα. Στην πάλη μα να σώσουμε ε, ανθρώπου, αποφασίσαμε να αγοράσουμε ένα σκάφο συλλέγοντα ε, δωρεέ το, από το GoFund. Και είμαστε περιορισμένοι. Ήταν σε ανοιχτή θάλασσα τα που βουλιάζαν τα πλοία και δεν έφταναν στην ακτή. Ακολουθήσαμε όλου του διάβλου έγκριση και ε, τελικά καταχωρήσαμε ε, στον ιολόγιο τα σκάφη μας. Τώρα ξαναζείτε τη στιγμή αυτή μαζί μα. Ήταν πρωινό τη 14η Ιανουαρίου, περίπου 2 ώρα το πρωί. Ήμουν στο αυτοκίνητό μου ε, περιπολώντα και μου είπε ένα από, από την ομάδα των εθελοντών ότι στην Νότια Ακτή βουλιαζε ένα σκάφο. Όμω δεν δόθηκαν συντεταγμένε. Αυτό σήμαινε ότι η κατάσταση από κακή γίνει χειρότερη. Ξέραμε ότι οι άνθρωποι αντιμετώπιζαν προβλήματα, δεν ξέραμε πού. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν στη θάλασσα και ίσω ότι μπορούσαν να έχουν μόνο λίγα λεπτά ζωή. Και ήξερα ότι δεν μπορούσα να αντέξω ξανά ε, να δω κάποιον να πνίγεται μπροστά μου ε, και ούτε να μπω στη θέση του να καταλάβω πως είναι να πνίγεσαι. Εγώ και άλλοι τέσσερις διασώστες ετοιμαστήκαμε αμέσω, πήγαμε στο λιμάνι και πήγαμε στο σκάφος διάσωσης και ξεκινήσαμε, ξανοιχτήκαμε για να σώσουμε αυτούς που ήταν στη βάρκα. Ειδοποίησαμε την ελληνική ακτοφυλακή που είπαμε να έρθουμε σε επαφή μαζί τους αν βρούμε το σκάφος ή την τοποθεσία του. Λοιπόν, έπλεα εκεί πέρα και προσπαθούσα να βρω το πλοίο που βούλιαζε. Ξαφνικά ένα στρατιωτικό, ένα πλοίο του πολεμικού ναυτικού έφτασε ε, με μεγάλη ταχύτητα και πριν να το καταλάβουμε σταμάτησε και συλληφθήκαμε. Το σκάφος που ήμασταν εκεί ήταν αυτό το ίδιο σκάφος που είχαμε χρησιμοποιήσει πριν 15 ώρες για να σώσουμε 51 ζωές με την άδεια των αρχών και τρέμω να σκεφτώ ποια θα ήταν η μοίρα αυτών των ανθρώπων εάν δεν είχαμε αυτό το σκάφο για να ξεκινήσουμε τη δουλειά μα. Είμαστε στο λιμάνι, στο γραφείο των αρχών, περίπου πέντε ώρε χωρί εξήγηση. Ζητήσαν πανελειμμένα να μιλήσουμε με τι πρεσβείε μα, αλλά συνέχισαν να μα αρνούνται αυτό το δικαίωμα. Σε 9 το πρωί, εγώ και οι άλλοι Δανείοι ε, θελοντέ ε, μα ζητήσαμε να πάμε στο γραφείο ανάκριση. Οι αξιωματικοί δεν μπορούσαν να μιλήσουν αγγλικά ο ανακριτή κάτι τύπωνε ναι, επί 10 λεπτά και μου ζήτησε να του εξηγήσω τι συνέβη. Εγώ μιλούσα και εκείνο ε, ε, δαχτυλογραφούσε. Το πρόβλημα ήταν δεν καταλάβαινε αγγλικά. Τι έγραφε λοιπόν στον υπολογιστή του. Αφού τελείωσα, μου έφερε ένα έγγραφο και μου είπαν το υπογράψω. Απάντησα ότι δεν υπογράφω τίποτα χωρί να έρθει ο δικηγόρο μου έδωσαν στους άλλους δανούς εθελοντές ε, το ίδιο έντυπο να υπογράψουν. Τους είπα να μην υπογράψουν τίποτα αν θέλουν ξαναδούν τα παιδιά τους και τις ε, γυναίκες τους. Με έσπρωξαν εκτός της έσανάκρισης και το ίδιο και τους Είδα τους άλλους και τους είπα να μην υπογράψουν πριν να μιλήσω με δικηγόρο ή πριν μιλήσω με την πρεσβεία. Τελικά, μετά από επανειλημμένες αποτυχημένες απόπειρες από τις λιμενικές αρχές, έπρεπε να έρθουν σε επαφή με τις πρεσβείες μας και τελικά βρήκαμε ένα δικηγόρο. Από ό,τι κατάλαβα, το έγγραφο που θέλαμε να υπογράψουμε έλεγε ότι ήμασταν στην Τουρκία διακινώντα ανθρώπου προ την Ελλάδα και είχαν πρόσφυγε στο σκάφο μα. Ψευδό κατηγορήθηκα για διακίνηση ανθρώπων, δεν υπήρχαν στοιχεία να το αποδείξουν αυτό. Αυτό διατείνομαι. Ήμουν στα ελληνικά ύδατα χωρί πρόσφυγε στο σκάφο μου. Άλλοι αρχέ πολύ γρήγορα το ξέχασαν αυτό. Πέρασα 48 ώρε στην κράτηση και μου πονάει το στομάχι μου σκεφτόμενο του 8 πρόσφυγε που πέθαναν τότε, γιατί εμεί ήμασταν φυλακισμένοι και δεν υπήρχαν άλλα δυσοστικά σκάφη στη θάλασσα. Μέχρι τώρα οι αρχέ. Δεν κατάλαβα γιατί ξοδεύτηκε τόση ενέργεια για να καταστρέψουν ζωέ σα ή να σώνονται αθώοι. 48 ώρε περάσαν στη φυλακή και μετά ο καθένα έπρεπε να ε, πληρώσει εγγύηση για να φύγει. 10.000 ε, ευρώ που πληρώσω. Μετά την απελευθέρωσή μου δεν με πετράπει να φύγω από την Ελλάδα για ένα χρόνο και 8 μήνε. Εν τω μεταξύ αυτό δεν με σταμάτησε τι ανθρωπιστικέ μου προσπάθειε και τα προγράμματά μου. Εξακολουθούσα να καταβάλω προσπάθειε ούτω ώστε πιστέτε πρόσφυγε να δίνω στέγαση, ε, ενδύματα, ανθρωπιστική βοήθεια, τρόφιμα. Δεν είχα κανένα σκάφο πια διότι είχε κατασκευθεί. Αυτή δεν με σταμάτησε, συνέχισα να διασώζω ανθρώπου. Καμιά φορά κολυμπούσα 300-400 μέτρα και μετά επέστρεφα με το σκάφο ε, ε, στο οποίο επέβαινε πρόσφυγε. Αφού σταμάτησα να φτάνω σε μεγάλου αριθμού στα ελληνικά νησιά ε, αυτά τα σκάφη, λόγω συμφωνία Ευρωπαϊκή Ενώση Τουρκία, πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα, ξεκινώντα και εφαρμόζοντα προγράμματα για βοήθεια στου πρόσφυγε. Και στι 16 Αυγούστου του 2017, μετά από ένα χρόνο και 8 μήνε, τελικά μπόρεσα να φύγω από την Ελλάδα και να επιστρέψω στην οικογένειά μου. Ακόμα εκκρεμούσαν οι κατηγορίε και έπρεπε μετά από 9 μήνε να δικαστώ, το Μάη, 7 Μαου του 2018. Παρά τις ε, ε, τις διάφορες κατηγορίες που δεν σταθούσαν για εννέα μήνες ε, η ζωή μου σταμάτησε και ήταν μεγάλη δυνατότητα ότι θα αντιμετώπιζα τελικά ε, την υπόλοιπη ζωή μου διαβίου κράτηση. Έχασα τα πάντα. Ε, σκεφτόμουν ποιο θα με απασχολήσει αν έχω μια ε, ισόβια καταδίκη στο κεφάλι μου. Ισόβια στη φυλακή γιατί, γιατί σώσα ζωέ, παιδιά από το να πνιγούν. Η μετανάστευση είναι ένα κοινό φαινόμενο για τη μήνα, για την περιοχή δηλαδή μέσα Ανατολή, Ανατολική Βορειοαφρική. Η Μεσόγειο είναι μια δό για τη μετανάστευση. Οι αντιλήψει γι' αυτό έχουν αλλάξει με την πάροδο του χρόνου ε, λόγω τη αλλαγή τη οικονομική και κοινωνική κατάσταση. Η περιοχή EU μήνα είναι μια περιοχή όπου πάντα κανονικά μορφή επικρατούσε. Η μετανάστευση συμβάλλει σημαντικά στη συνύπαρξη στην περιοχή. Σήμερα η Ευρώπη παλεύει με έναν γυράσκοντα πληθυσμό και χρειάζεται τους μετανάστες, αλλά η αδυναμία της Ευρώπης στο σύνολό τη να διαχειριστεί την ισχυρή πίεση των ροών προσφύγων προς Συρία, Ιράκ, Αφγανιστά και από άλλες συγκρούσεις, καθιστά πολύ δύσκολο το να βρει κανείς την αναγκαία ισορροπία και να διαχειριστεί ε, την αυξανόμενη πολιτική ξενοφοβία. Η κοινωνία των πολιτών πάντα ήταν ο πρώτο που ανταποκρινόταν στι κατερίγου καταστάσει ανθρωπιστικέ. Δεκάδε ε, αλληλεί, ε, δικηγόροι και άνθρωποι που ζούσαν στι νότιε ευρωπαϊκέ ακτέ έσωναν και υποστήριζαν πρόσφυγε και μετανάστε αντικαθιστώντα τι μη υφιστάμε κρατικέ δομέ. Και βλέπω ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την κρίση από μόνη της. Ανησυχητικέ εξελίξει όπω η σύλληψη τριών εθελοντών στη Λέσβο τον περασμένο μήνα δείχνουν ότι πιέζεται η κοινωνία των πολιτών και είναι θολή εικόνα, σκοτεινή εικόνα που διαγράφεται η την προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι ανθρωπιστέ αυτοί ε, αντιμετωπίζουν σοβαρέ κατηγορίε. Υπάρχει υποψία ότι είναι διακινητέ και κατασκοπία. Μία από αυτέ είναι η Σάρα Μαρντίνη, που θα θυμόσαστε. Ήταν η πρόσφυγα από τη Συρία που ε, το 2015 ε, σχεδόν πνίγηκε ε, όταν άρχισε να βουλιάζει το φουσκωτό τη. Ε, και, και η αδελφή της και η Σάρα ε, πήδησαν στη θάλασσα ενώ βούλιαζε και τρεις, επί τρεις ώρες κολυμπούσαν προς τη Λέσβο τραβώντας το σκάφος, σωθήκαν όλοι. Λοιπόν, αυτή και συνάδελφος ο Σιμ Μπάιντερ αφιέρωσε μήνες της ζωής του για να βοηθήσει τον κόσμο. Ήταν Βιετναμέζος πρόσφυγας ο πατέρας του που πήγε στη Γερμανία μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ. Σαν ήθελε να κάνει τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος και να μπορέσει να εκτελεί στα καθήκοντά του. Και ήθελα να το κάνει αυτό, κυρίε και κύριοι. Βλέπω ότι ο κόσμο ε, κραυγάζει για βοήθεια και αν άλλοι θέλουν να αποκριθούν στι φωνέ αυτέ, σα εκλυπαρώ να βοηθήσετε ανθρωπιστέ όπω είναι η Σάρα και ο Σον. Πιστεύω στην ανθρωπότητα και πιστεύω ότι υπάρχει πολλή ανθρωπιά σε αυτή την αίθουσα εδώ σήμερα και γι' αυτό σα παροτρύνω να μπείτε στη θέση μα και σκεφτείτε τι θα κάνατε αν σα κατηγορούσαν για κάτι που είναι εναντίον αυτού που πιστεύετε. Τι αν κάποιο έλεγε ότι όλοι σε αυτή την αίθουσα αντιπροσωπεύουν το κακό, ε, την απάτη, την ανηλικρίνεια. Έτσι αισθάνθηκα και εγώ όταν μου είπαν ότι θα μπορούσα να αντιμετωπίσω ισόβια στη φυλακή, διότι προσπαθούσα να βοηθήσω τον κόσμο. Τελικά απαλλάχθηκα από κατηγορίε και δεν πέρασα τι υπόλοιπε μέσα τη ζωή μου πίσω από τη, τα κάγκια τη φυλακή λόγω αυτών των ισχυρισμών. Αλλά υπάρχει, υπάρχουν άνθρωποι που αντιμετωπίζουν βάσει κατηγορίε και βοήθησαν αυτού που είχαν ανάγκη. Είναι μια διεθνή υποχρέωση να, εξαιρεθούν, να εξαιρεθεί ανθρωπιστική βοήθεια από την τιμωρία για να εξασφαλίσουμε την ισχύ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των θεμελιωδών θα πρέπει να υπογραμμιστεί ε, η νομοθεσία και πολιτική όταν βοηθούμε τους ανθρώπους και τους διασώζουμε. Και θα πρέπει και οι συνθήκες υποδοχές να βελτιωθούν. Και κοιό και ανεξάρτητοι θελοντές θα πρέπει να, αποτε... να προστατευτούν από ποινικοποίηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να μεταρρυθμίσει την υφιστάμενη νομοθεσία και να έχει ένα, μια πολιτική για άσυλο και μετανάστευση. Αυτό δεν συμβαίνει σε εν μία νυχτή. Και θελοτυφλώντας αυτούς που πνίγονται εντωμεταξύ δεν είναι η σωστή απάντηση. Θα ήταν παράνομο σύμφωνα με το διεθνέ δίκαιο με το διεθνέ δίκαιο, οποιοδήποτε σκάφο που είναι κοντά σε ένα άλλο και αντιμετωπίζει κίνδυνο πρέπει να βοηθηθεί ανεξάρτητα από τη σημαία του σκάφους ή που βουλιάζει. Εάν δεν βοηθήσει κανείς είναι έγκλημα ε, παράληψης. Μια μόνιμη ε, λύση χρειάζεται, μια μεταρρύθμιση που θα εξασφαλίζει ότι η αλληλεγγύη δεν είναι έγκλημα και ε, οι πρόσφυγες που δεν έχουν ταξιδετικά έγγραφα μετανάστες θα πρέπει να, έχουν, να χάνουν των βασικών δικαιωμάτων. Κυρίε και κύριοι, ταπεινώνω τον εαυτό μου Στεκόμενο μπροστά σα, σα παρακαλώ να βοηθήσετε του ανθρωπιστέ που αντιμετωπίζουν κατηγορίε μόνο και μόνο γιατί έχουν ιδεώδη και θέλουν να βοηθήσουν. Για την ανθρωπότητα. Από την καρδιά τη Ευρώπη, καλώ όλου αυτή την αίθουσα να δραστηριοποιηθούν, να εξασφαλίσουν ότι θα απελευθερωθούν από την κράτηση αμέσω. Δεν του αξίζει να αντιμετωπίζονται σαν εγκληματίε. Θέλω να ευχαριστήσω καθένα εθελεντή που έκανε θυσίε για του άλλου. Χωρί αυτού θα είχαμε μεγαλύτερη κατάρρευση στην Ευρώπη. Ευχαριστώ για τον χρόνο Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα αλλάζουμε ταχύτητα κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε μια παρουσίαση για το πώς τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν την οδηγία. Ζων Κρούν θα μας τα πει. αναπληρωτή διευθυντή μετανάστευση του Υπουργείου Ιστορικών τη Γαλλία. Θα μα πει πώ υλοποιείται η οδηγία περιδευκών στη Γαλλία. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. 10 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, σα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν μπορώ να μιλήσω εξ όλων των άλλων χωρών, θα μιλήσω εξ τη Γαλλία. Και θα πω κυρίω τη νομική σκοπιά Υπενθυμίσατε κύριε Πρόεδρε, όταν κάνετε την εισαγωγική σας παρέμβαση, και το είπαν και οι προλαλήσαντες ε, ε, μου ομιλητές, υπενθυμίσατε την ανθρώπινη διάσταση. Τα κράτη-μέλη δεν είναι τέρατα, την έχουν ε, υπόψη του στη διάσταση αυτή, Παρά παράτυπη μετανάστευση διαμέσου της Μεσογείου είναι και θέμα το οποίο πρέπει να προληφθεί. Πρέπει να καταπολεμηθούν ε, τα δίκτυα διακίνησης ε, εμπορίας ανθρώπων ε, ανάντι. Δεν είναι στόχος μας μόνο η καταστολή και επιβολή κυρώσεων στο πλαίσιο του ποινικού δικαίου. Για να μην ακρηγορήσω, δεν θα σας υπενθυμίσω την οδηγία του 2002, που είναι και θέμα της ημέρδας αυτής. Η Γαλλία μετέφερε στο Εθνικό Δίκαιο την οδηγία. Ήδη στο δίκαιο της χώρας προβλέπονταν κυρώσεις για όσους ε, βοηθούσαν κάποιους να εισέλθουν παράνομα στη Γαλλική επικράτεια. Προσαρμοστήκαμε όμως ε, με την ε, οδηγία το 2016 συγκεκριμένα. Δεν θέλω να επανέλθω στα φαινόμενα μετανάστευσης. Νομίζω ότι ο εκτελεστικός διευθυντής ε, της Frontex ε, που θα ακούσουμε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του στη συνέχεια θα τα πει καλύτερα από μένα και για τα κυκλώματα και για τις τεχνικές που χρησιμοποιούν ε, για την διακίνηση των μεταναστών. Άρα εγώ θα δω το νομικό ζήτημα και από την πλευρά της Γαλλίας. Σε ό,τι αφορά τη βοήθεια ε, για ξένους να μπουν και να διαμείνουν στην Γαλλική επικράτεια. Έχουμε στον ε, κώδικα περί αλλοδαπών ε, ένα άρθρο που ορίζει το ποινικό αδίκημα και ένα άλλο άρθρο που ορίζει τα μέτρα εξαίρεσης από δίωξη. Υπάρχουν και άρθρα για επιβαρυντικές επιπτώσεις, περιπτώσεις όταν ε, υπάρχει οργανωμένη ομάδα, συμμορία ή και για τις εξαιρέσεις που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ανθρωπιστική βοήθεια αλλά και την ε, οικογενειακή επανένωση μελών ε, οικογένειας μεταναστών. Άρα εδώ μιλάμε για οικογενειακή αλληλεγγύη και υπάρχει εξαίρεση. Σε ό,τι αφορά τα γεγονότα. Η Γαλλία δεν είναι στην πρώτη γραμμή σε ό,τι αφορά τη θαλάσσια μετανάστευση λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Δεν φτάνουν τα πλοία, τα σκάφη σε γαλλικά λιμάνια καταρχάς. Πάνε αλλού πριν οι άνθρωποι αυτοί. Βέβαια μας αφορά το θέμα της βοήθειας, ε, της διευκόλυνσης της εισόδου στη χώρα, της παράτυπης ε, μετανάστευσης, ιδίως γιατί από το 2015 Έχουμε επαναφέρει τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Η Γαλλία λοιπόν είναι αντικείμενο των λεγόμενων δευτερογενών ροών, όπως τις λέμε. Και έχουμε και ένα πολύ ιδιαίτερο φαινόμενο στο Καλέ. Από τη Βόρεια Θάλασσα που θέλουν να περάσουν μέσω του Καλέ στην Αγγλία μετανάστες. Ε, πέρυσι τώρα να σας πω κάποιοι. Το 2017 103.000 ε, άνθρωποι εντοπίστηκαν ε, σε κατάσταση παράτυπης μετανάστευσης ρεκόρ για τη Γαλλία σε ό,τι αφορά την πρόληψη και την καταπολέμηση της διακίνησης μεταναστών η γαλλική αστυνομία 330 κυκλώματα παράνομης εργασίας ε, και μετανάστευση 139 ήταν κυκλώματα που σχετίζονται με τη διευκόλυνση εισόδου στη χώρα. Οι γαλλικές αρχές, καστικές αρχές ε, για το 16 χωστιά, για το 17, μάλλον παρόμοια είναι. 764 καταδίκες ε, είχαμε 230 ε, μάλιστα ήταν ποινές φυλάκισης χωρίς αναστολή αρκετά σταθερό στα τελευταία χρόνια των καταδικών αλλά σε ό,τι αφορά τη σπινές κράτησης χωρίς αναστολή βλέπουμε αύξηση που σημαίνει ότι είναι όλο και πιο δομημένα, οργανωμένα και καλά εξοπλισμένα τα κυκλώματα. Σε ό,τι αφορά το νομοθετικό μηχανισμό που έχουμε στη διάθεσή μας. Είπε ένας προλαλήσοντας ε, κάτι για το Γαλλικό Σταγματικό Δικαστήριο που τον Ιούλιο απεφάνθη επί του θέματος σε ό,τι αφορά το άρθρο που σας προανέφερα, το άρθρο για τις εξαιρέσεις από δίωξη. Τι λέει το άρθρο αυτό. πριν παρέμπτω το σταγματικό συμβούλιο. Έλεγε ότι δεν μπορούσε να υπάρξει δίωξη αν το φυσικό ηθικό πρόσωπο δεν είχε κάποιο άμεσο ή έμεσο αντάλλαγμα και αν παρήχε νομικές συμβουλές, φιλοξενία, ιατρική βοήθεια, για να εξασφαλίσει αξιοπρεπή ε, συνθήκες, αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης στο άτομο που ήταν το αντικείμενο της βοήθειας. Άρα εμείς θεωρούσαμε ότι έχουμε σωστά μεταφέρει, το ίδιο κρίνει και η Κομισιόν, τη σχετική οδηγία. Το Σταματικό Συμβούλιο άσκησε κριτική σε αυτή τη διάταξη λέγοντας ότι όχι ότι δεν συνάδει με την οδηγία, αλλά με τη συνταγματική αρχή της αδελφοσύνης, της αδελφότητας. Φρατερνητέ. Και δύο είναι τα συμπεράσματα που αντλεί. Πρώτον, ότι πρέπει να προσθέσουμε στο δίκαιο το γαλλικό εξαίρεση για τη διευκόλυνση κυκλοφορίας και όχι μόνο εισόδου και διαμονής. Και το δεύτερο, ρητός πρέπει να εφαρμόσουμε την εξαίρεση που προβλέπεται όταν ο στόχος είναι αμυγός ανθρωπιστικός. Υπήρχε ένα νομοσχέδιο, το οποίο εκπονεί το τότε, και σε αυτό το νομοσχέδιο, που ήταν πιο γενικό ως προς τη θεματολογία του, συμπεριλάβαμε τις ε, σχετικές τροποποιήσεις για να καλύψουμε τα αιτήματα του Σταγματικού Συμβουλίου και έτσι το νέο κείμενο αυτού του γαλλικού νόμου που ορίζει τις εξαιρέσεις από δίωξη πλέον προβλέπει ότι δεν μπορεί να υπάρξει δίωξη φυσικού νομικού προσώπου όταν δεν υπάρχει άμεσο έμεσο αντάλλαγμα. Αυτό ήταν από την αρχή δεν. Και όταν συνίσταται στην παρχή νομικών συμβολών, δικαστικής πλαισίωσης, παροχή βοήθειας με αποκλειστικά ανθρωπιστικό στόχο. Είναι διάταξη δεν αναφέρει συγκεκριμένα ε, κάποιες περιπτώσεις, είναι πιο γενικόλογη, ε, είναι μια πιο γενική διάταξη που καλύπτει πολλές ενέργειες από τη στιγμή που ο στόχος τους είναι ανθρωπιστικός αμυγός. Θα ήθελα εδώ να αναφέρω δύο πράγματα για να διευκρινίσω κάποια πράγματα. Ότι κάποιες μη μας κατηγορούν ενίοτε ότι δεν εξαιρούμε τον κερδοσκοπικό χαρακτήρα στο άρθρο που κάνει λόγο για την αξιόπινη πραξία το αδίκημα. Για επιχειρησιακούς λόγους έγινε αυτό. Όταν μια υπηρεσία αστυνομική ξεκινάει τη δικαστική έρευνα, δύσκολα μπορεί να πει εκείνη τη στιγμή, τέλο πάντων δεν είναι πάντα εύκολο, να πει κατά πόσον υπήρξε, δεν υπήρχε αντάλλαγμα αν υπήρξε κέρδος δηλαδή. Και επειδή δεν είναι σίγουρο και επειδή υπάρχει αυτό στον ορισμό ε, της παράβασης, το ότι πρέπει να υπάρχει κερδοσκοπικός χαρακτήρας, πρέπει να υπάρχει αντάλλαγμα, δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν πολλές έρευνες. Άρα αυτό θα ερχόταν σε αντίθεση με το στόχο, τον ωφέλιμο στόχο της οδηγίας αυτής εξ αρχής. Η τα δίκτυα, τα κυκλώματα χρησιμοποιούν όλα και επιτεδευμένα μέσα για να μην υπάρχει παραδείγματος χάρη μια πληρωμή στο γαλλικό έδαφος, να μην φαίνεται ξεκάθαρα ε, τι γίνεται, υπάρχουν κάποιοι μεσάζοντες ε, και είναι πολύπλοκο το όλο σύστημα και όλος ο μηχανισμός που χρησιμοποιούν για να μπορούν να τους πιάσουν στο γαλλικό έδαφος. Έχουμε λοιπόν συνδυάσει τώρα δύο διαφορετικά άρθρα για το στόχο μας. Μια άλλη διευκρίνηση. Και με αυτήν θα ολοκληρώσω. Σε ό,τι αφορά την είσοδο. Η διευκόλυνση εισόδου δεν είναι αντικείμενο, πώς να το πω, μιας ρητής διάταξης στο γαλλικό δίκαιο για εξαίρεση από δίωξη για ανθρωπιστικούς λόγους ανθρωπιστικοί λόγοι μιλάνε, έχουν να κάνουν μόνο για την διευκόλυνση διανομής και το 2018 διευκόλυνση και της κυκλοφορίας. Ό,τι αφορά την διευκόλυνση εισόδου, υπάρχει μια διαφοροποίηση λοιπόν μεταχείρισης της εισόδου αφενός και της ε, ε, διαμονής ε, και κυκλοφορίας αφετέρου. Επικυρώνεται και από το Σταγματικό Συμβουλίο το 2018 Και αυτό αιτιολογείται ως εξή. Σε ό,τι αφορά την είσοδο. Αυτός που βοηθάει, που αρέχει βοήθεια, δεν βοηθάει απλά ε, τον παράτυπο μετανάστη, τον φέρνει μέσα στη γαλλική επικράτη και έτσι δημιουργεί, ε, παράγει, δημιουργεί γεννά την ε, παράτυπη αυτή κατάσταση. να περάσει τα σύνορα δηλαδή ο μετανάστης για να είναι παράτυπος τα χερσαία σύνορα κυρίως. Πρέπει να περάσει τα ισπανικά, βελγικά κτλ σύνορα. Αν ένας που είναι στο Ιταλικό-Βελγικό σύνορ, ε, ένας μετανάστης ε, που είναι σε κακή κατάσταση, μπορεί εκεί να του παράσχει κάποιος βοήθεια, αλλά να μην τον περάσει ε, απέναντι στα γαλλικά σύνομα, του παράσχει στην Ιταλία, στο Βέλγιο, βοήθεια στην Ιταλία κτλ. Εκεί που αντιμετωπίζει το πρόβλημα, την ανάγκη. Αυτά σε ό,τι αφορά τη διευκόλυνση εισόδου. Δεν υπάρχει λοιπόν διάταξη. Ε, είναι μια γενική αρχή του ποινικού δικαίου, γιατί για το ποινικό δίκαιο μιλάμε εδώ, που λέει η γενική διάταξη, ότι η κύρωση υπάρχει αν υπάρχει πρόθεση στα πεπραγμένα. Και υπάρχει και η ανάγκη. Ε, αν δηλαδή ε, υπήρξε ανάγκη να γίνει κάτι. Αν Δηλαδή ήταν ανάγκη να σωθεί ένας άνθρωπος. αλλά δεν το αναφέρουμε αυτό συγκεκριμένα με συγκεκριμένη διάταξη στη, στα, στο άρθρο για τη διευκόλυνση εισόδου. Είπα λοιπόν ότι έγινε η τροποποίηση του νόμου και με την τελευταία αυτή τροποποίηση νομίζουμε ότι η νομοθεσία μας πλέον συνάδει πλήρως με τη στάση και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμμορφούνται προς αυτή, αυτές τις συστάσεις, είναι απόλυτα ισορροπημένοι, πιστεύουν νομοθεσία αφενός μεταξύ ανάγκης καταστολής, ε, της διευκόλυνσης εισόδου διαμονής και της δράσης των κυκλωμάτων διακίνησης και αφετέρου της δράσης των ανθρωπιστών. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάμε στις δύο τελευταίες ε, παρεμβάσεις ε, σύντομες. Πριν περάσουμε στην συζήτηση, έχουμε ένα σύντομο ηχογραφημένο μήνυμα του κυρίου Λετζέρη, εκτελεστικού διευθυντή της Frontex, ο οποίος κολλείεται ε, και για να είμαι δίκαιος έρχεται εδώ αρκετά συχνά ε, οπότε για να είμαστε δικοί μαζί του σήμερα έχει κόλλημα έστειλε όμως ένα ηχογραφημένο μήνυμα ευτυχώς είναι μόνο 5 λεπτά αλλά τα τελευταία δύο λεπτά φορούν το, το θέμα μας. Πάμε λοιπόν. Είναι τιμή και ευχαρίστησή μου να μιλώ στην Επιτροπή σας ε, ως επικεφαλής της Frontex με τις επιχειρήσεις της ε, στα εξωτερικά σύνορα ε, τις επιχειρήσεις Οι άνθρωποι της Frontex ε, συχνά είναι οι πρώτοι οι οποίοι βλέπουν τα θύματα διακίνησης όταν φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως δεν γνωρίζετε το ότι η Frontex έχει βοηθήσει στην διάσωση σχεδόν 23.000 ανθρώπων μέχρι στιγμής φέτος. Επίσης υπάρχουν και επιχειρήσεις διάσωσης ε, οι οποίες είναι υπό τον έλεγχο και διοίκηση των εκάστοτε κρατών μελών. Μετά την αποβίβαση ακολουθεί ταυτοποίηση, καταγραφή και έλεγχος παρατύπων μεταναστών. Μαζί με τις εθνικές συνοριακές αρχές της χώρας άφηξης, η υπηρεσία μας κατόπιν παραπέμπει τα άτομα στις αρμόδιες αρχές. Με τον τρόπο αυτόν, όσοι θέλουν να ζητήσουν άσυλο κατευθύνονται στις αρχές ασύλου. Πιθανά θύματα διακίνησης παραπέμπονται στην αστυνομία που ίσως τους παραπέμψουν σε διεθνείς ή τοπικές ΜΚΟ. Ασυνόδευτοι ανήλικοι παραπέμπονται στην αρχή προστασίας ε, ανηλίκων και οι έγκυες γυναίκες ε, παραπέμπονται στα τοπικά κέντρα υγείας διεθνείς οργανισμοί, όπως η Πατήρμοστια του ΙΕ και ο Διεθνής Οργανισμός για τη Μετανάστευση, εμπλέκονται σε πολλές από αυτές τις παραπομπές, όπως επίσης και πολλές τοπικές εμικιό, μεταξύ των οποίων και ο Ερυθρός Σταυρός και το Save the Children. Όμως, δεν είναι μόνο μέσω αυτών των επιχειρήσεων που εμπλέκεται η Frontex. Από το 2011 η Frontex παρέχει εκπαίδευση και οικοδόμηση δυνατοτήτων σε κράτη-μέλη και τρίτες χώρες για την καταπολέμηση της διακίνησης ανθρώπων και την αύξηση της προστασίας των παιδιών. Μάλιστα, έχουμε αφιερώσει ένα ολόκληρο έργο για να βοηθήσουμε τους συνοριοφύλακες να ανοιχνεύουν τα ανήλικα θύματα διακίνησης και σωματεμπορίας. Η υπηρεσία άρα Ε, εξακολουθεί να δουλεύει αδιάκοπα με τα κρατη για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των εξωτερικών συνόρων. Ο ρόλος μας ε, για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος δεν σημαίνει ότι παραμελούμε την διάσωση ζωών εν πλώ, σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από τις διεθνείς υποχρεώσεις μας. Δεν υπάρχει κάποια αντίφαση, κατά την άποψή μας, με το να δείχνουμε ανθρωπιά στο θύμα και να συνεισφέρουμε αφενός και στην καταπολέμηση του εγκλήματος. Στόχο έχουμε να διατηρήσουμε την ασφάλεια της ευρωπαϊκής επικράτειας με την προστασία των εξωτερικών συνόρων και με το να καταπολεμούμε το οργανωμένο διεθνές έγκλημα. Η υπηρεσία μαζί με τους ε, συνεταίρους της ε, στη Europol και τη Eurojust παίζει έναν σημαντικό ρόλο σε τομείς όπως η καταπολέμηση της διακίνησης ανθρώπων, λάθροδιακίνηση μεταναστών, διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, απάτη ειδικών φόρων κατανάλωσης κλπ. Ένα σημαντικό στοιχείο λοιπόν της εντολής μας είναι ακριβώς η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τα οποία κατόπιν μοιραζόμαστε με τη Europol και τα κράτη-μέλη για τον στόχο ποινικών ερευνών με τον τρόπο αυτό στηρίζουμε τις εθνικές αρχές στην εφαρμογή της οδηγίας περί διευκόλυνσης. Κυρίε και κύριοι βουλευτές, ως μια νέα υπηρεσία η Frontex δεν μετέχει στις πολιτικές συζητήσεις για την αναθεώρηση της σχετικής οδηγίας. Η μεταφορά της οδηγίας βεβαίως είναι στα χέρια των κρατών μελών και η ανεξάρτητη δικαιοσύνη της κάθε χώρας θα κρίνει το εάν έχει λάβει χώρα διευκόλυνση σε κάθε συγκεκριμένο περιστατικό. Κλείνοντας όμως, θα ήθελα να υπογραμμίσω το γεγονός όλοι μας, ε, η Frontex, τα κράτη-μέλη, οι ανθρωπιστικές ε, μήκυο, έχουμε στόχο να δώσουμε βοήθεια στα θύματα κατά την άφηξή τους και στο να μειωθεί ο αριθμός των θυμάτων τους επόμενους μήνες και χρόνια. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ. Oh, Μάλιστα. Τώρα ε, ε, αυτά μας πατρονάρουν αυτές οι βλακίες εδώ πέρα. Δηλαδή, εντάξει, ο εκτελεστικός διευθυντής ε, ήθελε να κάνει δήλωση αντί να στείλει κάποιον, από την άλλη τώρα βλέπουμε βίντεο next time we don't um, Αλλά έρχεται αρκετά συχνά. Και βεβαίω ε, είναι σε επαφή για αυτό το ζήτημα. Οπότε ε, το, ας μην έχουμε ε, ηχογραφημένα μηνύματα σε αυτό το πνεύμα. και μια που έχουν μείνει μόνο δύο βουλευτές ε, θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν. Ξέρω ότι έχετε 10 λεπτά, έχετε προετοιμάσει ομιλία, αλλά αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε εδώ είναι η οδηγία και οι κατευθυντήριες γραμμές. Μπορείτε να μας στείλετε τις κατευθυντήριες γραμμές. Αν δεν ξέρετε πότε θα τις λάβουμε, εντάξει. Αν δεν τις λάβουμε, κάντε μας μια ανάλυση του που θεωρείτε ότι βρισκόμαστε. Ξέρω ότι μπορείτε να μιλήσετε 10 λεπτά για τη Μεσόγειο λοιπά... Αλλά ας το εστιάσουμε λίγο. Δηλαδή, 5 λεπτά για να μην μου φύγουν και οι τελευταίοι βουλευτές. 10 λεπτά άμα θέλετε εντάξει, αλλά θα προτιμούσα 5. Και ε, αν δεν πρόσεχαν ε, το θέμα είναι να δούμε τις κατευθυντήριες γραμμές κομισιών, γιατί ρεαλιστικά δεν θα υπάρξει αναθεώρηση της οδηγίας. Ο κόσμος πεθαίνει, θέλουμε να κάνουμε κάτι, θέλουμε να παρέμβουμε. Πρέπει να κάνουμε κι εμείς ε, να πούμε κάτι ως Κοινοβούλιο, έτσι. Οπότε, ζητήσαμε από την Κομισιόν να κάνει κάτι. Έχετε λοιπόν κάποια εμπειρία, έχετε ξανάρθει εδώ, να είστε λίγο στιασμένους. Try and uh, focus on this point and welcome. Thank you, Chair. And, uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κατευθείαν στο θέμα. Μετά από τις χειρότατες αυτές παρουσιάσεις που ακούσαμε και την παρέμβαση του κυρίου Διευθυντού της Frontex και την πολύτιμη συνεισφορά του εκπροσώπου της γαλλικής κυβερνήσεως που παρουσίασε τη θέση ενός κράτους μέλους. Δεν είχαμε κατά το παρελθόν κάτι τέτοιο σε άλλες συζητήσεις και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Μου ζητήσατε να είμαι συγκεκριμένο. Λοιπόν, κατευθυντήριες γραμμές. Αναφέρονται στο ψήφισμά σας που θετήσατε τον Ιούλιο φέτος. Ποιο είναι το θέμα. Από την αξιολόγηση της οδηγίας το 2017 δεν ήταν ε, το ερωτηματικό, δεν ήταν θέμα χρονισμού, αλλά κατά πόσο ήταν σχετική η οδηγία με το πρόβλημα και τι αντίκτυπο έχει. Οι κατευθυντήριες γραμμές, η άλλη νομοθετική φύσεως παρέμβαση της οδηγίας θα παραγάγει αποτελέσματα. Τα ευκταία. Κάναμε ανάλυση αξιολογώντα την οδηγία. Και ακολούθησαν και άλλε αναλύσεις. Όλα αυτά που κάναμε δεν άλλαξαν το συμπέρασμα της περσινής αξιολόγησης. Με νομοθετική παρέμβαση, με κατευθυντήριες γραμμές, δεν θα βρούμε μακροπρόθεσμη λύση που θέλουμε όλοι. Για να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική τραγωδία που αντιμετωπίζουμε όλοι και που τρέμουμε. και υπάρχει έλλειψη συστημικής λύσεως για τη μεταναστευτική, ε, το μεταναστευτικό πρόβλημα. Δύο στοιχεία τονίσαμε στην αξιολόγηση που ίσχυαν πέρσι και φέτος. Πρώτον, ακόμα και όταν υπάρχουν σε εθνική νομοθεσία εξαιρέσει ανθρωπιστική βοήθεια και υπάρχουν στα κράτη-μέλη της Frontex αυτές οι προβλέψεις, εξακολουθούν να συμβαίνουν αυτά που ακούσαμε. Κανένα νομοθετικό μέτρο, ούτε οδηγία, ούτε προσανατολισμοί έχουν το ευκταίο αποτέλεσμα. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, το είχαμε αναφέρει στην αξιολόγησή μας και αυτό. Δεν υπήρχαν αρκετά στοιχεία, τουλάχιστον αυτό ίσχυε το 2017. Δεν είχαμε στοιχεία να ξέρουμε προς ποια κατεύθυνση να κινηθούμε. Τώρα αυτό αλλάζει μετά το 2017. Σαν αποτέλεσμα αυτού φέτος ξεκινήσαμε μια διαδικασία. Καλέσαμε όλους τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών που έχουν στοιχεία και διαδραματίζουν ένα ρόλο στο συγκεκριμένο θέμα να μας δίνουν στοιχεία. Ποικίλουν οι καταστάσεις από έρευνα και διάσωση στη Μεσόγειο και φτάνουμε στις περιστάσεις που αναφέρθηκαν από τη Γαλλία. οι διαστάσεις είναι διαφορετικές ανάλογα με το κράτος μέλος. Είναι και θέμα στάσης έναντι των ΜΚΟ εν γέννη. Υπάρχει επικοινομορφία δράσεων και πραγματικότητας. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν κατανοητά και να καταγραφούν για να επιλέξουμε την καλύτερη λύση. Όπως είπα, ξεκίνησε η διαδικασία. Φέτος το Μάιο έγινε η πρώτη συνεδρίαση. Θα γίνει και άλλη περιμένουμε και την άποψη των φορέων της κοινωνίας των πολιτών. Είμαστε επαφή μαζί τους. Τους προσφέραμε τη δυνατότητα να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα, να υπάρχει διάδραση με τους εκπροσώπους κυβερνήσεων των κρατών μελών εκείνων που είναι στην άλλη όψη του νομίσματος. Λόγω των λύσεων που βρίσκονται λύση περισσότερο στην εθνική νομοθεσία ή πώς εφαρμόζεται αυτή η νομοθεσία στα εθνικά δικαστήρια ή στις αγγελίες, πιστεύουμε ότι αυτή η διάδραση η στις εισαγγελιε πιστευουμε φορέων κοινωνία των πολιτών και εθνικών αρχών είναι πάρα πολύ σημαντική. Προσφέραμε τέτοια πλατφόρμα συζητήσεων. Θέλουμε να συλλέξουμε τα στοιχεία, περισσότερα από αυτά που είχαμε μέχρι τώρα. Να δούμε ότι υπάρχει προθυμία από αυτού του φορείς να συμμετάσχουν σε αυτή την πλατφόρμα που πρότεινα. Δύο άλλα πράγματα που υπενοήθησαν, αλλά δεν αναφέρθησαν από τις παρουσιάσει των συναδέλφων. Σαφώς. Να έχουμε το εξή υπόψη. Έχουμε αυτές τις ιστορίες, τις πραγματικές τη ζωή που ακούσαμε, που μα συγκλώνησαν και ρίχνουν την διάσταση της ανθρώπινης τραγωδίας. μου ότι εκατοντάδε χιλιάδε ζωές σώθηκαν τα τελευταία δύο-τρία χρόνια λόγω της δράσης που ανελήφθη. Να το έχουμε υπόψη και αυτό. Αναφέρθηκαν νόμιμοι οδοί. Δεν είναι τόσες πολλές οι λύσεις όπως θα θέλαμε και τόσο αποτελεσματικές. Τώρα περισσότερες άδειες διαμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκδόθηκαν από ό,τι κατά το παρελθόν και έχουμε και αναλήψει υποχρεώσεων η μετεγκατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερες παρά ποτέ. Μικρό βήμα, δεν αρκεί αυτό. Εάν θέλουμε μακροπρόθεσμες λύσεις, αυτές προέρχονται από νομοθετικής φύσεως προτάσεις που υποβάλαμε, το πακέτο ε, που υποβάλαμε εδώ και δύο-τρία χρόνια. Τα τελευταία δύο χρόνια συμπληρώναμε τις προτάσεις. Και όπως ξέρετε, καλύτερα από μένα, έχουν κολλήσει. Εάν προχωρήσουν τα νομοθετική φύσεως μέτρα, τότε μακροπρόθεσμα θα βρεθεί η λύση που χρειάζεται. Καλύτερο αυτό παρά οι προσανατολισμοί. Δεν τι απορρίπτουμε τι κατευθυντήριε γραμμέ. Θα υποβάλουμε ένα έγγραφο, θα συλλέξουμε το κατάλληλο υλικό, αλλά κατά την άποψή μα η λύση θα προέλθει από την υιοθέτηση του πακέτου. Έχουμε ένα πρόγραμμα μετεγκατάσταση, ένα σύστημα προστασία των ετούντων άσυλο, ισχυρότερο ε, ισχυρότερη υπηρεσία για το άσυλο. Όλα αυτά είναι στο πακέτο και αν υιοθετηθούν όλα αυτά θα είμαστε σε καλύτερη θέση. Ευχαριστώ κύριε Τεράτσι για αυτά που είπατε. Πρέπει να εξετάσουμε όλα αυτά τα θέματα. Μείνετε εκεί που είστε για να συζητήσουμε. Να το θέσω αυτό και α μην είναι ρεαλιστικό και α είναι αφελέ. Θέλω να το εκφράσω όμω να βρούμε μια λύση μέχρι τώρα της θητεία. Είναι δραστηριοποιημένοι οι συνάδελφοι οι δύο που είναι εδώ, οι δύο κυρίες. Ας ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Μπάρμπαρα Σπινέλη πρώτη. Και μετά η Μαρή Κριστίν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εν πρώτη να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας τον κύριο Νέστλερ και τον ιδρυτή της Humanity των Σαλάμ Αλτίν. Η μάχη τους είναι και δική μου. Να ευχαριστήσω και τους συντάκτες της μελέτης Fit for Purpose, τις δύο ε, συν, ε, συγγραφείς της μελέτης. Άκουσα αυτά που είπε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιστεύω ότι μια αναδιατύπωση οδηγίας είναι κάτι απαραίτητο. Νέοι προσανατολισμοί χρειάζονται. Το είπαμε και εμείς στο ψήφισμά μας. Ίσως αυτό μακροπρόθεσμα να μην επιλύσει το πρόβλημα. Βραχυπρόθεσμα όμως πρέπει να κινηθούμε και βραχυπρόθεσμα η ΜΚΟ και διάφορες ενώσεις ποινικοποιούνται. Χρειάζονται νέοι προσανατολισμοί και αυτό το λέω επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και κυρίως η οδηγία διευκόλυνσης προφανώς αντιτίθεται με αυτά που λέει ο ΟΗΕ, κυρίως από το Smuggling Protocol, άρθρο 16.3. Εκεί η βοήθεια, η παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολία και ιδιαίτερος στους undocumented migrants, στους μετανάστες χωρίς αξιδιωτικά έγγραφα είναι κάτι υποχρεωτικό. Ενώ στην οδηγία δεν είναι κάτι υποχρεωτικό, αλλά εθελοντικά παρέχεται από τα κράτη-μέλη. Άρα αυτό είναι κάτι πολύ απαραίτητο. Να πω κάτι άλλο, πιο θεμελιώδες. Αντιμετωπίζουμε σε διάφορες χώρες, ξεκινώντας από τη χώρα μου, την Ιταλία, μια πολιτική στρατηγική συγκεκριμένη εξωτε, εξωτερήκευσης της πολιτικής ασύλου και από την εξωτερήκευση δημιουργούνται τα προβλήματα που συζητούμε. Ποινικοποίηση ή ασδήποτε δραστηριότητας έρευνας και διάσωσης παροχής βοήθειας προς μετανάστες χωρίς τα ταξιδιτικά έγγραφα στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Το λέω αυτό δίνοντας το παράδειγμα της Ιταλίας. Αντιμετωπίζουν μια κλιμάκωση. Πριν, πρώτα ξεκίνησε η ποινικοποίηση των σκαφών των ΜΚΟ και άρχισε να διάζει από θάλασσα, από σκάφη που έδιναν βοήθεια. Τα αποκαλούσαν ταξί μεταναστών σαν οι μετανάστες ήταν άνθρωποι που πάνε σε θάλασσα αναψυχής στη Μεσόγειο, στις ακτές για αναψυχή. Η κλίμακωση συνέχισε με το εξή. Ποινικοποιήθηκαν και στατιωτικά σκάφη Ιταλικά του πολεμικού ναυτικού. Την, στο σκάφος Διτσιώτη. Άρα υπάρχει εσωτερική σύγκρουση εντός των φορέων του Ιταλικού κράτους. Η πολιτική εξωτερήκευσης τη διαχείριση των συνόρων γίνεται σε αντίθεση με πρακτικές που ακολουθούν τα σκάφη του πολεμικού ναυτικού της Ιταλίας αλλά και το Υπουργείο Αμήνης της Ιταλίας και αυτό με ανησυχεί πάρα πολύ στην περίπτωση της Ιταλίας προβλέπεται και ένα νέο διάταγμα για την ανάστευση και την ασφάλεια όπου όλες οι κατηγορίες συναθρίζονται οι μετανάστες χωρίς έγγραφα, μετανάστες μετά έγγραφα, οι τρομοκράτες, οι διακινητές, οι smugglers. Όλοι θεωρούνται επικίνδυνα άτομα που θα μπορούσαν να χάσουν την Ιταλική υπηκότητα εάν κάνουν το παραμικρό, την παραμικρή παράβαση. Έχουμε ένα όραμα δηλαδή της ηθαγένειας που είναι μονοεθνική για πρώτη φορά με τα πολεμικά. Και όλα αυτά τα πράγματα, κατά την άποψή μου, είναι μια πολιτική στρατηγική. Δεν χρειάζεται νέος προσανατολισμός. Είναι μια ε, μινιμαλιστική προσέγγιση αυτή απλώς των νέων προσανατολισμών. Δεν αρκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπάρμπαρα. Κοιτώντας εδώ πέρα το ψήφισμα, το φετινό, το οποίο μιλάει για τις κατευθυντήριες γραμμές κτλ., και την ε, ολοκληρωτική προσέγγιση της μετανάστευσης. Ε, βεβαίως ε, το καιρό εκείνο, το 2016, που λέει ότι θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται η αρχή ότι όσοι έχουν ανάγκη δεν θα πρέπει να ποινικοποιούνται κτλ. Και τώρα πλέον έχει νερωθεί εντελώς. Αλλά Ε, είναι προφανές το ότι θέλαμε τότε. Απλά λέω το τι συνέβη. Αυτό συνέβη. Ε, συγγνώμη, έτσι έγιναν τα πράγματα. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν είναι ερώτηση. Ε, άποψη εκφέρω, μου επιτρέπετε. Μαρή Κριστίν, πες και εσύ κάτι και μετά θα επανέλθει το πάνελ να πούνε και άλλα πράγματα. Σε ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους πρώτους τέσσερις ομιλητές γιατί έριξαν φως κατά κάποιο τρόπο στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επιβεβαίωσαν τις δικές μας ανησυχίες και τις δικές μας προσδοκίες ό,τι αφορά τη μεταφορά της οδηγίας για τη διευκόλυνση στο εθνικό δίκαιο. Πιστεύω ότι περισσότεροι εδώ στο Ευρωκοινοβουλίο πιστεύουμε ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει σύγχυση μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθησας, ανθρωπιστικής αλληλεγγύης και διακίνησης ανθρώπων. Επίσης θα ήθελα να πω ότι η ανεπάρκεια πόρων, ιδίω ό,τι αφορά τη διάσωση στη θάλασσα, μετά το Μαρενόστρομ Νόστρομ και τη σχετική απόφαση, τι οδήγησαν όλα αυτά. Να έχουμε αυτή την κατάσταση στη Μεσόγειο, την ανήκουστη κατάσταση που βιώνουμε σήμερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζουμε εδώ ότι γίνονται οι και υπάρχει διάσωση στη θάλασσα από όταν προέκυψε καινούργια δεδομένα στην Ιταλία που σώζονται οι άνθρωποι. Ε, ακούμε ότι υπάρχει ένα σκάφος μια ΜΚΟ. Σώζονται από τους επίσημους οργανισμούς ποτέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση τόσοι άνθρωποι και τα κρατημέρια. Πού πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Θα ήταν ενδιαφέρον να το μάθουμε αυτό. Να έχουμε απαντήσει. Και γιατί τόση κινδυνολογία. Όταν υπάρξει ένα σκάφος ε, με 55 ή 58 συγκεκριμένα άτομα ΜΚΟ δεν ξέρω και εγώ πόσε μέρε πέρασαν ε, για να δεχτεί κάποιο κράτος μέλο να δεχτεί 55 άτομα. Όνειδο ντροπή για τα κράτη-μέλη της Ένωσης που δεν μπορούν να υποδεχθούν ένα σκάφο και βάζω και τη Γαλλία κύριε Ντεκρόν μέσα. Εντάξει, δεν είμαστε στην πρώτη γραμμή, αλλά δεν είμαστε όπω η Δανία, έτσι. Και είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από την Ισπανία. Και η Ισπανία άνοιξε τι πόρτε τη. Η Γαλλία δεν τι άνοιξε και το σκάφος ε, που το δέχτηκαν ε, στην Ισπανία πέρασε από τα νυχτά της Κορσικής. Και νομίζω θα ήταν πιο απλό να σταματήσει στην ε, Κορσική και να μην φτάσει μέχρι τη Βαρκελόν. Μην υπερβάλλουμε σε αυτά που λέμε. Δεν την αφορά το θέμα τη Γαλλία, τόσο δεν την αφορά που δεν ζήτησε καν σε αντίθεση με αυτά που είπατε, την αποκατάσταση των συνόρων για την μετανάστευση, αλλά για την τρομοκρατία το ζήτησε. Και εμείς εδώ αγωνιζόμαστε και θέλουμε διευκρινήσεις για το θέμα αυτό. Δεν υπήρξε μεταναστευτική ροή μεταξύ Ιταλίας και Γαλλίας. Υπάρχει απλή άρνηση της Γαλλίας να εφαρμόσει το Διεθνές Δίκαιο, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και το Εθνικό Δίκαιο. Και ο νομάρχης ε, των Αλπ Μαριτήμα πολλές φορές έχει καταδικαστεί γιατί δεν σέβεται τα δίκαια αυτά που προανέφερα. Πείτε μου ό,τι θέλετε, αλλά δώστε μου και συγκεκριμένα στοιχεία για την εφαρμογή της νομοθεσίας και του δικαίου. Δεν εφαρμόσετε το δίκαιο. Λοιπόν, να πω και κάτι ακόμη. Έχω κάποιες αμφιβολίες. Αφού έχουμε εκπρόσωπο των γαλλικών αρχών και μας μίλησε για τη μεταφορά της απόφασης του Συνταγματικού Συμβουλίου στο γαλλικό δίκαιο δράτω με τις ευκαιρίες για να εκφράσω τις αμφιβολίες που έχω για το πόσο συνεπής είναι αυτή η νέα νομοθεσία και με τη συνταγματική αρχή περί αδελφοσύνης που αναγνωρίζει και το Συνταγματικό Συμβούλιο. Πράγματι, έχουμε το τρίτο εδάφιο αυτού του άθρου 624, αλλά δεν καταλαβαίνω. Το είπανε και πολλοί ΜΚΟ στην γαλλική κυβέρνηση. Παραμένει το θέμα της άμεσης ή έμεσης συνδρομής, διευκόλυνσης. Δεν κατάλαβα εσεί τι σχέση ε, κάνατε μεταξύ αυτού του κερδοσκοπικού ανταλλάγματος, του κέρδους αφενός και της άμεση ή έμεση συνδρομής. Δεν είναι το ίδιο και το αυτό. Παρ' όλα αυτά, εσείς, όχι εσείς προσωπικά, η γαλλική κυβέρνηση, οι γαλλικέ αρχές, προσθέσατε κάτι το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην απόφαση του Συνταγματικού Συμβουλίου. όρος στρικτεμό μανιτέρη, είπατε αυστηρός, αμυγός. Δεν λέει αυτό ε, η απόφαση της Κομισιόν μιλάει για ανθρωπιστικό χαρακτήρα και εσείς μιλάτε για αμυγός, για αυστηρά ανθρωπιστικό χαρακτήρα. Στρίκτε μα. Έχουμε διγαλικά δικαστήρια. Χωρίς να θέσω υποαμφισβήτηση την γαλλική δικαιοσύνη εν γέννη, την εμπιστεύομαι. Το είδαμε και την απόφαση του Σταματικού Συμβουλίου. Αλλά υπάρχουν κάποια δικαστήρια που τόλμησαν να πούν ότι υπήρξε έμεση διευκόλυνση, έμεση συνδρομή, διότι ήταν, λέει, ακτιβιστές που καταδικάστηκαν και ότι είχαν όφελος. Μα πού οδεύουμε, πού πάμε εξ αρχής, επειδή ποτέ έχουν ένα όφελος, έχουν, θέλουν, έχουν συμφέρον να βοηθήσουν ανθρώπους που είναι ε, σε δύσκολη θέση από ανθρωπιστική και μόνο ε, συνείδηση και αλληλεγγύη, λέτε ότι αυτοί οι άνθρωποι παρήχαν διευκόλυνση. Μήπως αφήνουμε πάρα πολλά περιθώρια τελικά ερμηνεία. για αυτή την καταραμένη την έννοια, ανθρωπιστικό στόχος. Και τελευταίο, Με εξέπληξε αυτό που άκουσα να λέει ο εκπρόσωπο τη Κομισιόν, που κάνει ένα παραλληλισμό μεταξύ των ζώων που σώζονται. Συμφωνούμε όλοι βέβαια ότι σώζονται ζωέ, αλλά αυτό που μα ανησυχεί, και το είπε, όχι μόνο ένα πολύ ομιλητές, είναι η αναλογία των θανάτων ε, σε σχέση με τις διελεύσεις. Αυξάνει το αριθμό σε αυτών που πεθαίνουν. Κάτι δεν πάει καλά επομένως. Γιατί δεν πάει κάτι καλά, ακριβώς γιατί δεν υπάρχει νόμιμη είσοδο δεν υπάρχει νόμιμη οδός. Αν υπάρχει, υπάρχει λόγο εθνικότητας. Μην τα βάλουμε σε τσουβάλι. Ρεκόρ μιλήσατε στις άδειε διαμονής. Ποιες τις παίρνουνε. Για δείτε τη χώρα. Δεν έχει ρυθμιστεί το ζήτημα της Μεσογείου ούτε των διελεύσεων. Πρέπει να ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι. Μη μας σχετίζετε την κατάσταση στη Μεσόγειο με τον αριθμό αδειών παραμονής. Δεν ξέρω τι ισχύει με τα νούμερα του 17, αλλά σε ό,τι αφορά το 16, οι Ουκρανοί ε, στην Πολωνία ήταν, ε, στη μερίδα, είχαν τη μερίδα του λαού Τι σχέση έχει αυτό με τη Μεσόγειο. Ευχαριστώ. Τέλος, η Άννα Γκόμης. Ναι. Και εγώ. Εγώ άλλωστε έχω δηλώσει δημοσίως ε, στη χώρα μου ότι ζητάω από την κυβέρνηση της Πορτογαλίας ε, να εγγράψουμε στο νιολόγιο το Aquarius και τα άλλα πλοία που πλέον δεν βρίσκουν νιολόγιο. Έτσι θα σώσουμε την αξιοπρέπειά μας. Όποιος δεν το καταλαβαίνει δεν αξίζει να δουλεύει ε, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιλαμβάνομαι ότι οι ε, κατευθυντήριες γραμμές δεν προσθέτουν τίποτα ε, όσον αφορά τις υποχρεώσεις μας στο πλαίσιο της συνθήκης και διεθνών συνθήκων. Και απορώ που και κάποιες κυβερνήσεις που δεν είναι φασίστες και ρατσίστες ακολουθούν τη ρητορική τους, ε, του Σαβίνη και του Όρμπαν και λένε ότι οι ΜΚΟ που μόνο ζωές ε, σώζουν ε, θα μπορούσαν ε, να ποινικοποιηθούν ως ε, διακίνητες. Μάλιστα, οι κυβερνήσεις αυτές με το να μην ανοίγουν ασφαλείς και νόμιμες ε, διόδους για, προσφυγές και, για πρόσφυγες και τούντες άσυλο τρέφουν τα δίκτυα, την πίσνα αυτή που τροφοδοτεί τα δίκτυα των ε, διακινητών και σωματεμπόρων. Δεν είναι η ανθρωπιστική παγίδα δηλαδή, είναι η παγίδα της business. Και με το να μην παρέχουν νόμιμες και ασφαλείς διόδους, πράγματι επιτρέπουν στους διακινητές να είναι οι διαχειριστές των ροών αυτών. Όπως και ο κύριος Γκουτιέρες είπε όταν ήταν ε, ε αρμοστής για τις πρόσφυγες. Γι' αυτό λοιπόν ε, μου έρχεται αναγούλα όταν ακούω αυτά τα πράγματα για το κατά πόσο η επιστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ή δεν είναι αυτή. Σας παρακαλώ λοιπόν κύριοι Γιούνκερ, Μογκερίνη, Αβραμόπουλε, πείτε στις κυβερνήσεις ποια είναι η ανθρωπιστική και νομική τους υποχρέωση να σώζουν ζωές και να οργανώσουν μάλιστα τις ροές προσφύγων και μεταναστών για να μην συνεχίσουν να ισχυροποιούν τη μαφία των διακινητών. Και, επί τη ευκαιρία, πρέπει να προσευχήσουμε την προσοχή στο ότι δεν ασχολούνται με τους πλούσιους αλλοδαπούς που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή έχουν λεφτά και πληρώνουν τις χρυσές βίζες, που είναι ένα σύστημα για να οργανωθεί η εισαγωγή οργανωμένου εγκλήματος. Εκεί πέρα δεν του πειράζει. Μάλιστα, μάλιστα. Να επανέλθουμε τώρα στους ομιλητές. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω. Λοιπόν, μία ερώτηση προς τον κύριο Νέστλερ και τον κύριο Σαλάμ Αλντίν. Ε, έτσι σύντομα, αν μου επιτρέπετε. Μία γρήγορη απάντηση στις ερωτήσεις της Μπάρμπαρα Σπινέλη, της κυρίας Βερζιά. Ε, και της Άννας Γκόμες, δεν ξέρω, έφυγε. Ξέρετε την πολιτική κατάσταση, τα είπε η κυρία Σπινέλη. Βλέπετε την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, πώς είναι η κατάσταση από τη σκοπιά των ΜΚΟ τη δική σας σκοπιά που προσπαθείτε να βοηθήσετε και πώς βλέπετε το άμεσο μέλλον ε, ημών και άλλων ανθρωπιστών που θέλουν να βοηθήσουν. Έτσι μια ιδέα δώστε μας ε, για να κλείσουμε. Έχοντας αυτά λοιπόν κατά νου, έτσι από τα αριστερά προς τα δεξιά, πείτε μας ε, δύο και ο καθένας το πολύ παρακαλώ. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να πάνε και στα σπίτια τους διερμηνείς. ξεκινήσουμε λοιπόν από τον δόκτορα Νέσλερ και να ακούσουμε τους υπόλοιπους. Πείτε μας λοιπόν ένα τελευταίο σχόλιο. Ευχαριστώ. Να σας πω, ε, έχουμε μεγάλη απογοήτευση. Και εμεί ε, ήμασταν σίγουροι ότι κάνοντα αυτή τη δουλειά υπό το φω των όσων συμβαίνουν, Εμείς σώζουμε ανθρώπους που πνίγονται και προσπαθούμε να φτιάξουμε μια ασφαλή δίωδο προς την Ευρώπη. Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες δεν, ε, για να μην αναγκάζονται να παίρνουν ε, το δρόμο αυτό που κινδυνεύουν. και φοβόμαστε ότι τελικά η Ευρώπη θα πάει σε ένα μοντέλο Αυστραλίας όπου δεν θα υπάρχει τρόπος να μπει κανείς και ε, θα έχουμε κλειστά σύνορα. Οπότε βλέπουμε το πώς συζητιέται δημοσίως το τελευταίο χρόνο σαν να είναι μια αρρώστια ή κάποιοι να προσπαθούν να κατακτήσουν την Ευρώπη. Και εμείς τους έχουμε δει κατά πρόσωπο να παλεύουν και πραγματικά είναι απογοητευτικό να βλέπουμε πώς διαμορφώνεται η δημοσία συζήτηση. και το νομοθετικό πλαίσιο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε και εμείς για τη δουλειά που κάνετε. Ευχαριστούμε και τους συναδέλφους σας στις διάφορες ΜΚΟ για το ανθρωπιστικό σας έργο. Περί αυτού πρόκειται, περί ανθρωπιστικής προσπάθειας. Ευχαριστώ. And I hope we don't go to the Australian model, but it's very telling that έτσι αισθάνεστε ότι πάμε προς το αυστραλιανό μοντέλο. Το ένστικτό σας ήθελα να ακούσω τι σας λέει. Πρόθεσή μας δεν είναι να φέρουμε αξιωματούχους από κράτη-μέλη να ακουστούν. Θέλουμε και μόνο. Θέλουμε ισορροπημένο πάνελ. Υπόθηκαν κάποια πράγματα στα οποία θα να απαντήσετε ίσως κύριε Ντεκρίν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στο γενικό ερώτημα του πάνελ να απαντήσω. Πώς βλέπουμε τα πράγματα εν συνεχεία. Προφανώς, οι διακινητές όταν φέρνουν τους ανθρώπους με στα βαρκάκια στα λιβικά, στα όρια των λιβικών υδάτων και μετά με κινητό τηλέφωνο ειδοποιούν τις ΜΚΟ ή την Ιταλική ακτοφυλακή για να λάβουν τα άτομα, δεν είναι κανονική κατάσταση. Δεν πρέπει να διαρκέσει αυτό. Η λύση δεν ξέρω που είναι. Αυτό που κάνουν οι ΜΚΟ είναι μια διάσωση. Κάτι πολύ σημαντικό. Τους ο φόρο τιμής. Πρέπει να βρούμε και τα αίτια του φαινομόνου. με αυτό ασχολούνται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κάτι μερή, είτε πολυμερό είτε διμερό σε συνεργασία με τις χώρες Αφρικής, στις χώρες της παράκτιες, με το Μαλί, τον Ήγυρα, με τις χώρες του Σαχέλ, έγινε συνήθω κορυφή της Βαλέτας, ακολούθησαν και άλλε πρωτοβουλίε. έγινε μια προσπάθεια να σταματήσει αυτή η ροή που κατευθύνεται προς τη Μεσόγειο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. όσον αφορά αυτό που μας απασχολεί σήμερα το απόγευμα. Ο τρόπος των προβλεπωμένων κυρώσεων για τη βοήθεια εισόδου διαμονής των αλλοδαπών. Σημερίζομαι κάπως την ανάλυση του κύριου Ντοράτσα. Μπορούμε να βελτιώσουμε τη σύνταξη του ποινικού μα κώδικα. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε αυτό, δεν μιλώ για τι άλλε χώρε. Να επιφέρουμε βελτιώσει που είναι στο περιθώριο όμω. Ο τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται τα κείμενα το σημαντικό. Όπω εφαρμόζεται η οδηγία. Μπορούμε να τη βελτιώσουμε. Και το εθνικό δίκαιο των χωρών. Πρέπει η εφαρμογή των κειμένων τα δικαστήρια να είναι ομοιογενής και να συνάδει με το πνεύμα των ισιών των κανόνων και κειμένων. Δεν ξέρω αν έχω χρόνο να απαντήσω την κυρία Βερζιά. Δεν θέλω να αρχίσει όμως γαλογαλικός διάλογος. Κοιτάξτε, πολύ γρήγορα. Κάνα δίλεπτο έχουμε έτσι άλλους συναδέλφους. Τελευταίο σχόλιο παρακαλώ. Πάνω σε αυτό που είπε η κυρία Βερζιά. Η θέση της Γαλλίας όσον αφορά τα σκάφη στην Μεσόγειο. Εφαρμόζουμε το δίκαιο των θαλασσών. Η αποδοχή στο πρώτο ασφαλή λιμένα αυτού του σκάφους είναι κάτι που πρέπει να ισχύει και μετά είναι θέμα αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό που συνέβη για τους 58 που μιλήσατε για τα Aquarius έγινε με συμφωνία μεταξύ των τεσσάρων χωρών, εμβαλωματική λύση κλπ. Πρέπει να κινηθούμε προς καλύτερη διοργάνωση της αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Κύριε Τεντεράτς, από εδώ και πέρα τι κάνουμε. Ευχαριστώ. Σύντομα. Όπως είπε και ο πρόεδρος Γιούνκερ πρόσφατα, θα χρησιμοποιήσω τα λόγια για να δώσω κάποιες απαντήσεις σε αυτά που υπόθηκαν. Τι είπε ο κύριος Γιούνκερ. Ότι ο ίδιος δεν πίστευε ότι παλεύοντας να βρούμε μια λύση για 50 ανθρώπους σήμερα και άλλη λύση αύριο για άλλους 50, ότι έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα. Όσον αφορά τη μετανάστευση. Χρειαζόμαστε δομημένες λύσεις και για την αλληλεγγύη, σωστά αναφέρθηκε από τον Γάλλο συνάδελφο. Αυτό πιστεύουμε ότι θα δώσει τις αναγκαίες λύσεις. Παρά να προσπαθούμε να αναλύουμε και να χτενίζουμε τον ορισμό του αδικήματος. Υπάρχει σαφής ορισμός για τη διακίνηση, η διακίνηση ανθρώπων ποια είναι και υπάρχει και ορισμός ποια είναι η ανθρωπιστική βοήθεια. Οι ορισμοί υπάρχουν. Το πώ ερμηνεύουν τι διατάξει του ορισμού στα δικαστήρια. Αυτό αφορά τα δικαστήρια και τη δικαιοδοσία του. και εναρμόνιση αυτών, αυτό είναι κάτι που γίνεται σε εθνικό επίπεδο. Θέλουμε, πια, αυτή είναι η ιδέα, να αποφύγουμε φορεί τη κοινωνία των πολιτών να φτάνουν σε αυτή την κατάσταση και μόνο παρέχοντα τι λύσει που έχουμε εμεί στο πακέτο θα βρούμε άκρη. Ελπίζουμε ότι οι συνομοθέτες μέσω αυτού, δίνοντας χρόνο, και θεσμική ισχύ θα βρεθεί και η λύση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Θα πάω στον κύριο Αλντίν. Σύντομα, αφού σας ευχαριστήσω για τη δουλειά σας, ε, ξέρω ότι δεν είναι εύκολο, θα σας παρακαλούσα έτσι συνοπτικά να πείτε δύο-τρία λόγια μόνο. Θέλω σταματήσει αυτή η τρέλα. Να πάω να ποινικοποιούνται οι εργαζόμενοι στον ανθρωπιστικό κλάδο. Ο Σόν, η Σάρα, είναι στι φυλακέ. Ένα μήνα και δέκα μέρε ήδη. Λόγω κάποιων πολιτικών που λένε άμα τους βάλουμε στη φυλακή, τι, δεν θα έρχονται πρόσφυγες στην Ελλάδα. Εγώ ξέρω πόσο δύσκολο είναι. να σε κατηγορούν για κάτι τόσο τεράστιο. ώστε να την πληρώσεις μένοντας στους τους στη φυλακή. Όλοι θέλω να αναλάβουν δράση για την άμεσα απελευθέρωση από τη φυλακή. Να ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ. Εκτιμούμε ιδιαίτερα το έργο που κάνει και εσύ και οι φίλοι σου και οι άλλοι συναδελφοί σου. Ευχαριστώ πολύ. Η τελευταία λέξη στις δύο συναδέλφους που μας έβαλαν στο πλαίσιο. Θέλετε να πείτε κάτι για το άμεσο μέλλον. Σύντομα όμως. Πολύ γρήγορα πέντε. Πρώτον. Δεν αφορά μόνο τη Μεσόγειο το θέμα. Το ακούσαμε και στη συζήτηση αφορά τα χερσαία σύνορα της Ένωσης, την κατάσταση των διαμενόντων που αντιμετωπίζουν όλο και πιο εχθρική ε, αντιμετώπιση, συμπεριφορά το παράτυπα διαμένοντες. Σίγουρα ε, όλοι συγκινούμαστε από αυτά που συμβαίνουν στη Μεσόγειο, δεν είναι όμως ε, το μόνο μέρος όπου έχουμε επαναλαμβάνουμε τέτοια περιστατικά. Το δεύτερο, αποδοτικότητα του προπολογισμού. Προπολογισμό για τον έλεγχο των συνόρων τριπλάσιος σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. 34,9 δισεκατομμύρια αγγλικές λίρες. Πόσα θα πάνε για να μπαίνουν στη φυλακή άνθρωποι, πόσα θα πάνε για την καταπολέμηση της ε, ε, παράτυπης μετανάστευσης, της διακίνησης, ε, πόσα θα πάνε για την παροχή σχολικής εκπαίδευσης ε, στα, σε αυτά τα παιδιά. Λιγότερα δίνονται για τη διάσωση ανθρώπων, για αυτά που κάνει ο Αλντίν. 71 έχασαν τη ζωή του το 2015 σε ένα φορτηγό στην Αυστρία. Δεν είναι μόνο τα σύνορα της θάλασσας. Είχαν περάσει τρία διαφορετικά κράτη μετά την Ουγγαρία. Και τους έβλεπαν, τους παρακολουθούσαν, ε, τα κράτη-μέλη επέκλεπαν τις ενομιλίες τους. Εμείς έχουμε μιλήσει, η Λίνα και εγώ, με ανθρώπους που είχαν πρόσβαση πληροφορίες, που τους ακούγανε να λένε οι μετανάστες πεθαίνουμε, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Επειδή δεν υπάρχει διεθνή συνεργασία δεν έγινε τίποτα και πέθαναν αυτοί οι 71 άνθρωποι. Πώ θα αξιοποιήσουμε λοιπόν αυτά τα χρήματα, αυτό είναι το θέμα, για να καταπολεμήσουμε τη διακίνηση και να σώσουμε ζωέ και να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα. Διαβάστε την έκθεση παρακαλώ, τον Οκτώβριο θα δημοσιοποιηθεί και θα έχουμε και ένα βιβλίο σύντομα με πολύ περισσότερες λεπτομέρειες, μελέτη περιπτώσεων και διευκρινήσεις. Ευχαριστώ. Η Λίνα. Ακούγοντας ε, την συζήτηση αυτή σκέφτομαι ότι ε, η παράνομη διακίνηση μεταναστών είναι η νέα τρομοκρατία και πλέον δεν υπάρχουν ε, δικαιώματα ούτε ποινική δικονομία ε, για να παταχθεί απλά το θέμα αυτό το οποίο συχνά είναι πολιτικό. Και όπως βλέπουμε στα δικαστήρια ε, και οι διώξεις ε, πολιτικοποιήθηκαν, τα έγραφαν τα ΜΜΕ και τα λοιπά και υποτίθεται ότι αυτά θα τα έκριναν οι ανεξάρτητοι δικαστές όμως βλέπουμε μια πιστοχώρηση του κράτους ε, δικαίου και πόσο πιθανό είναι οι υποθέσεις αυτές ε, να μην ε, οδηγηθούν σε μια κατάσταση σαν την Ουγγαρία και σε άλλες χώρες. Οπότε εγείρεται ένα ευρύτερο θέμα κράτους δικαίου και το πού βρίσκεται το θέμα της παράνομης διακίνησης αυτή τη στιγμή είναι πολύ ψηλά στην πολιτική ατζέντα και όλοι θέλουν να προσφέρουν τις λύσεις τους ε, είτε τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα είτε όχι. Για πρέπει να είναι σαφές ότι δεν υπάρχει κάποια εξισορρόπηση ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διαχείρισης ε, συνόρων. Πρέπει να σεβαστούμε τα θεμελιώδη δικαιώματα και αυτό το λέει ξεκάθαρα ο κώδικας Σέγγεν και οι άλλοι κανονισμοί που έχει εγκρίνει και το Ευρωκοινοβούλιο και χαιρόμαστε που ε, είμαστε παρόντες και στις συζητήσεις της ε, Κομισιόν γιατί υπάρχει σοβαρή ανησυχία για το τι συμβαίνει στις επιχειρήσεις της ε, Frontex. Η επιχείρηση αυτή τη στιγμή άλλαξε όνομα από Ποσειδών σε Θέμης δεν έχει δικαίωμα αυτόματης αποβίβασης των όσων διασώζει στην Ιταλία. Οπότε έχουμε μία οπισθοχώρηση, έχουμε περισσότερη αβεβαιότητα. Οπότε βλέπουμε ότι ο παράγων που προσελκύει ακριβώς είναι ε, αυτός ο εκφοβισμός που ζει η κοινωνία των πολιτών. Δηλαδή το να μας λένε ότι εμείς ε, προσελκύουμε χωρίς να υπάρχουν κάποια σχετικά στοιχεία είτε μιλάμε για τη Μεσόγειο είτε για διανομή τροφίμων ε, στο συνδρομικό σταθμό του Παρισίων ε, δηλαδή αυτά τα πράγματα παραβιάζουν τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών όπως παραδείγματος χάρη το τεκμήριο της αθότητας ε, συχνά ακούμε ότι η παράνομη διακίνηση είναι ε, μεγάλη εγκληματικότητα και τόσα λεφτά διακινούνται και κερδίζουν πολλά οι διακινητές. Γιατί υπάρχει λοιπόν τόσο μεγάλη αντίσταση ε, όσον αφορά σε αυτό το κριτήριο περί ε, πραγματικού ωφέλου. Δηλαδή αν υπάρχει κάτι τέτοιο αργά ή γρήγορα η αστυνομία θα το βρει. Αλλά τον πιάνουμε αυτούς που χωρίς λεφτά λένε πού μπορεί κανείς να πάρει το λεωφορείο είναι και διασπάθηση δημοσίου χρήματος και σπατάλη αυτά. Για τη συνεργασία με τις ε, τρίτες ε, χώρες ε, είναι πολύ ανησυχητικό το ότι είχαμε ακούσει κάποιες περιπτώσεις αλλά ταυτόχρονα όταν πηγαίνει κανείς εκεί παραδείγματος χάρη η οργάνωση Jugendrettet έχει κάποια έχει ερευνηθεί για διακίνηση ενώ απλά διέσωζε κόσμο και η πίστα Μπουσουράη που μετέδιδε μηνύματα στην Ιταλική ακτοφυλακή ενώ η Ιταλική κυβέρνηση δωροδοκούσε τους ε, Λίβιους για να κρατήσουν εκεί πέρα τους μετανάστες και πρόσφυγες για να μην φύγουν από τη Λιβύη. Αυτό δεν ήταν ζήτημα παρά το ότι αυτή η παραστρατιωτική η Αλαμού και η Αλτασάντα τους θεωρεί ο ΟΗΕ το Γραφείο Εγκλήματος και Ναρκωτικών επίσης ως διακίνητες ε, είναι σε επίσημο κατάλογο και ξέρετε κάτι δεν πάει καλά δηλαδή έχουμε φύγει πλέον από την ανεκδοτολογία και τις ε, περιπτώσεις Έχει λήξει το ωραίο μας, σας αποχαιρετούμε